sono stato autorevolmente sollecitato. Με κάλεσε ένας πολύ σημαντικός ε, συνάδελφος να ξεκινήσουμε αμέσως τις εργασίες μας. Λοιπόν, έγκριση της, του σχεδίου ημερήσια διάταξη. Ε, ενημερωμένη εκδοχή τη ημερήσια διάταξη σα έχει αποσταλεί χθε. Προβλέπεται ένα νέο σημείο στην ημερήσια διάταξη, δηλαδή η παρουσίαση από πλευρά του Επιτρόπου Φούλε της ανακοίνωση για την αναθεώρηση της πολιτική γυπνίαση. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει κάποιο ψηλό προβληματάκι στην μετάφραση γιατί αλλάζουν οι γλώσσες από γαλλικά σε αγγλικά στην, ίδιο, στην ίδια καμπίνα. Μπορείτε να το ελέγξετε. Μάλιστα. Πρώτο σημείο είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης, επαναλαμβάνει ο Πρόεδρος. Έχουμε μία ενημερωμένη εκδοχή, η οποία σας παρουσιάστηκε χτες. Εντάξει, λύθηκε το θέμα. L'approbation de l'ordre du jour. Non, È il francese che sovrappone all'inglese, quindi non c'è inglese. I think the French translation was on the wrong channel. Μα νομίζω πως έχασε το δρόμο η γαλλική μετάφραση. I can show off and... Μπορώ να σας κάνω επίδειξη και να προσπαθήσω να μιλήσω αγγλικά, αλλά θα το μετανιώσετε. good now. Is that? For the French is good. Chiedi alla cabina inglese di parlare ε, ε, Ζητώ από την αγγλική ε, καμπίνα να ανάψει το μικρόφωνο της και να μιλήσει για να δούμε αν λειτουργεί. Ωραία, εντάξει, τακτοποιήθηκε το θέμα. Α πάμε πίσω. Έγκριση τη ημερήσια διάταξη πρώτο σημείο. Ενημερωμένη εκδοχή τη ημερήσια διάταξη, σας ε, δόθη εχθέ, σα εστάλει και προβλέπεται ένα νέο σημείο, η παρουσίαση από πλευρά του Επιτρόπου Φίλε τη ανακοίνωση για την αναθεώρηση τη πολιτική γυμνίαση και την ακύρωση της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών Υποθέσεων της Ισλανδίας λόγω των υφεστιακών υποθέσεών του. Άμα δεν υπάρχουν αντιρρήσει, εγκρίνεται. Δεύτερο σημείο, η έγκριση των πρακτικών τη συνεδρίαση τη 12η, 13η Απριλίου 2011 και τη συνεδρίαση 19 και 20 Απριλίου 2011. Δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Αυτά τα δύο πρακτικά εγκρίνονται. Τρίτο σημείο. Εδώ αντικαθιστώ τον πρόεδρο Αλμπερτίνη που χρειάστηκε να μείνει στην Ιταλία λόγω σημαντικών του πολιτικών υποχρεώσεων και που εκφράζεται λύπη του που δεν μπορεί να παραβρεθεί στη συνεδρίασή μας. Ελπίζω να σταθώ στο ύψος του Προέδρου Αλμπερτίνη. Σας ενημερώνω ότι η συνεδρίαση της 8 Σεπτεμβρίου ακυρώθηκε και θα αντικατασταθεί από μια συνεδρίαση τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο. Τέταρτο σημείο, η... μια αντιπροσωπεία έξι μελών της Επιτροπής ΑΦΕΤ πήγε στο Ουσμπεκιστάν 26 και 27 Απριλίου 2011. Αυτή η αντιπροσωπεία στη συνέχεια προσθέθηκε και ενώθηκε με την ομάδα οκτώ βουλευτών που ήταν από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Τουρκμενιστάν ε, και πήγαν στο Ουσβεκιστάν. Η κυρία Γκόμε ηγήθηκε αυτή τη αντιπροσωπεία στο Τουρκμενιστάν και οι δύο ομάδε ηγήθηκαν του κυρίου, ε, ηγήθηκε μάλλον των δύο ομάδων ο κύριο Βόμποντα που αντικατέστησε τον κύριο Μπαρτολότσι από την αντιπροσωπεία για την Κεντρική Ασία. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στους συναδέλφους Γκόμες και Σβόμποντα για να μας παραθέσουν τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια των δύο αυτών επισκέψεων. Θα ξεκινήσω με τη συνάδελφο Γκόμες. I Uh, θα, ήθελα να σας αναφέρω ε, τα όσα είναι στην επίσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Ουσβεκιστάν. Η βασική, το βασικό συμπέρασμα των μελών που επισκέφθηκαν το Ουσβεκιστάν είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια χώρα που χρειάζεται να επενδύσουμε σε με δική μας εμπλοκή ε, συμμετοχή και όχι απομόνωση παρά τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή και ιδιαίτερα στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπου είναι πολύ άσχημα τα πράγματα στο Ουσμπεκιστάν. Είναι πολύ ευρύτατα διαδεδομένη η παιδική εργασία και σχεδόν αποτελεί κρατική πολιτική Ε, συζητήσαμε τα θέματα με τους ε, ε, εκπροσώπους του Ουσμπεκιστάν δεν προσπάθησαν να, διαφύγουν, να ξεφύγουν από τη συζήτηση. Βέβαια είχαν ορισμένες διαφορετικές απόψεις, μάλιστα ορισμένοι προσπάθησαν να αρνηθούν την ύπαρξη του προβλήματος παιδικής εργασίας. Αυτό προσπάθησε να κάνει ένας βουλευτής, αλλά Το συζητήσαμε το θέμα και φυσικά προσπάθησαν ε, να μας ε, τονίσουν τα δικά μας μειονεκτήματα, τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα το οποίο βεβαίως ε, δεν μας προκάλεσε κανένα πρόβλημα, γιατί τονίσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη στον εντοπισμό προβλημάτων όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να πω, όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εμεί θίξαμε συγκεκριμένε περιπτώσεις και μετά από την επίσκεψη μαζί με την ε, Χάιδη Αουτάλα, ζήτησα από τον πρέσβη του Ουσμπικιστάν να αναγράψει τις περιπτώσεις ε, ε, φυλακισμένων κρατούμενων και μάλιστα ανταποκρίθηκε πολύ γρήγορα και μας έδωσε και γραπτή απάντηση. Εγώ αναλύω αυτές, αναλύω αυτές τις ε, πληροφορίες που λάβαμε, αλλά θα ήθελα να σημειωθεί ότι όντως αυτή η ενέργεια από πλευρά του πρέσβη δείχνει μια προθυμία την οποία διαπιστώσαμε και στο Ουσβεκιστάν για ε, συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάπως διαφορετικά δηλαδή είναι τα πράγματα από ό,τι στο παρελθόν. Συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ε, ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όπως είπα αναφέραμε την σφαγή του Αντιζάν, την ανάγκη για διεθνή έρευνα της υπόθεσης. Η επίσημη θέση είναι ότι έχει κλείσει το θέμα αλλά οι συνεδριάσεις που κάναμε, οι συναντήσεις που είχαμε με κάποιους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ε, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών είπαν εκεί ότι δεν θα υπάρξει πραγματική πρόοδος εάν συνεχίσουμε να αναφέρουμε το αντιζάν, καλύτερα να εστιάσουμε σε άλλα σημαντικά ζητήματα ε, που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης διαπιστώσαμε ότι το Ουσμπεκιστάν που γνωρίζει πολύ καλά την κεντρική του θέση στην Κεντρική Ασία ότι είναι η πιο πολυπληθής χώρα με σημαντική ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά και ούτω καθεξής ε, προσπαθεί μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λύσει τα προβλήματα που είναι βασικά, περιφερειακά. Ο, κυρίως το πρόβλημα του νερού που έχει τεράστιες επιπτώσεις για το Ουσμπικιστάν και για ολόκληρη την περιοχή. Και φυσικά ως προς αυτό θεωρήσαμε ότι οι Ουσμπέκοι ενδιαφέρονται για να τους βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με τους γείτονές τους λόγω των προβλημάτων αυτονομίας νερού που έχουν όλες οι χώρες περιοχής. Ως προς αυτό λοιπόν και σε σχέση με τους γείτονές τους επέκριναν κάπως το γεγονός ότι τίνουμε να εξετάζουμε την περιοχή αυτή ως ένα σύνολο, ενώ εκείνοι θα ήθελαν και όσον αφορά την, κατα... την κατανομή χρημάτων για τη συνεργασία, να έχουμε διαφορετική, διαφοροποιημένη μάλλον προσέγγιση, πρότειναν ότι κατά κάποιο τρόπο ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθά να δημιουργηθεί τεχνητά η ηγεσία στο Καζακστάν μέσω της ε, βοήθειας συνεργασίας κτλ. Το θέμα της παιδικής εργασίας είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ωστόσο, όπου πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να σημάνει τη διαφορά. Τόσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όσο και για άλλα θέματα. Πρόκειται για την ε, γεωργική μεταρρύθμιση, γιατί η παιδική εργασία συνδέεται ε, άρρηκτα με την συγκομιδή βαμβα... βαμβακιού. Απαιτείται πολύ χειρονακτική εργασία. Και αυτό οφείλεται στις αρχαϊκές μεθόδους ε, γεωργίας που χρησιμοποιούν στο βαμβάκι. Φυσικά αναφέραμε και άλλες περιπτώσεις για με συγκεκριμένα στοιχεία το βασικό θέμα της ελευθερίας της ενημέρωσης ούτως ώστε οι δικέ μας επαφές να είναι σε οποιοδήποτε τομέα και στον τεχνικό όπου υπάρχει μέγα ενδιαφέρον για τη συνεργασία με την Ένωση Υπάρχει ένα πρόγραμμα Tempus, το οποίο εκτιμάται όλος ιδιαίτερος, αλλά οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών διαμαρτυρήθηκαν ότι πολύ λίγες πληροφορίες παίρνουν για το πρόγραμμα αυτό και πολύ λιγοστές είναι οι ευκαιρίες για τους Ουσμπέκους πολίτες να συμμετέχουν. Διαμαρτυρήθηκαν και τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση του Ουσμπεκιστάν ε, ερευνά και συμπεριφέρεται με ιδιαίτερο τρόπο στους φοιτητές που φοιτούν στο εξωτερικό. Δεν μπορέσαμε βέβαια να έρθουμε σε επαφή με όλους όσους θέλαμε, γιατί είχαμε κάποια προβλήματα επικοινωνίας. Δεν καταλάβαμε ακριβώς βέβαια πού οφειλόταν και πολλοί άνθρωποι δεν μπόρεσαν να έρθουν. Δεν ξέρω αν σε κάποιο βαθμό θα αισθάνονταν εκτεθειμένοι ή ότι κινδύνευαν. Βέβαια, το θέμα του να συνυπογράψει την σύμβαση άρχου στο Ουσμπεκιστάν που έχει τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις αλλά και όσον αφορά δημοκρατικές διαδικασίες προτάθηκε από την ε, διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να, να πιέσουμε γι' αυτό και φυσικά προωθήθηκαν και διάφορες άλλες δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Ορισμένοι θεώρησαν ότι ε, μεγάλο τμήμα της εργασίας αυτής ε, οφείλεται στην Ευρώπη. Θεωρήθηκε σημαντική η δουλειά των οικονομικών μεταναστών του Ουσμπεκιστάν στη Ρωσία που προκύπτουν ως, αναδύονται μάλλον ως ε, ασκούντες πίεση για προτεσταντικές αλλαγές. Δεν μπορούμε να οριστολογούμε εκεί βέβαια, δεν μπορούμε να γενικεύουμε και να κάνουμε ένα διάλογο κενό περιεχομένου. Πρέπει να επιμείνουμε για συγκεκριμένες περιπτώσεις ε, έχουμε επαφές που να είναι υπόλογες στο Ουσμπεκιστάν ώστε να κάνουμε τη δουλειά που θέλουμε να κάνουν ιδιαίτερα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί και να αντιστοιχούν στο αίτημα των πολιτών εκεί ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί πιο δραστήρια και να βοηθήσει να λυθούν πολλά άλλα προβλήματα που όντω μπορούν να βρουν ε, λύση μόνο μέσω της περιφερειακής συνεργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκόμες. Το, συνα... το λόγο έχει ο κύριος Βόμποντα, παρακαλώ. Uh- Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι εκτιμώ τη δουλειά όλων των συναδέλφων που συμμετείχαν στην προσωπία. Ιδιαίτερο την Άννα Κόμες, από την Επιτροπή Εκτορικών Υποθέσεων, αλλά και την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή και επικοδομητική επίσκεψη. Αυτό που είπε η Άννα τώρα είναι θεωρώ απαράδεκτο εκ μέρους μας το ότι θέλουμε αέριο, πετρέλαιο, ανθρώπινα δικαιώματα, πρόοδο προς τη δημοκρατία από τις χώρες αυτές, αλλά δεν συμμετέχουμε με αντιπροσωπείες, μόνο με τον οίκο της Ευρώπης. Καλή δουλειά κάνουμε, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι αποδεκτό το έργο μας. Κατά δεύτερον, ο Επίτροπος Φίλε θα μας παρουσιάσει την ε, σχετική έκθεση δεν έχουμε όμως αντιπροσωπεία ακόμη εκεί. Άρα στις χώρες αυτές θέλουμε ε, ευρωπαϊκή παρουσία, ευρωπαϊκή δέσμευση. Αυτό μας βρίσκει όλους σύμφωνους. Η διαφορά τώρα στο Ουσπεκιστάν και στην διαδικασία ανοίγματο στο Τουρκμενιστάν είναι πιο διστακτική η όλη διαδικασία. Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα γιατί το γνωρίζουμε και εμείς και αυτοί ότι δεν είναι όλα εντάξει, αλλά χρειαζόμαστε έναν διάλογο ο οποίος έχει ξεκινήσει. Ελπίζουμε να συνεχιστεί και να διευρυνθεί. Η συζήτηση στο Κοινοβούλιο δεν ήταν πραγματική συζήτηση, ήταν μια παρουσίαση από την άλλη πλευρά και μια συζήτηση εκ μέρους μας. Είναι δύσκολα τα πράγματα με τον Υπουργό Εξωτερικών. Ήταν ε, μακρά η συζήτηση και πιο σκληρή και από τις δύο πλευρές. Φιλική μεν, αλλά σκληρή. Και φυσικά ξέρουμε ότι κι άλλοι παρακολουθούν την συνάντηση και ότι, θα πρέπει, ότι έπρεπε ο Υπουργός Εξωτερικών να ανταποκριθεί και σε τις ανάγκες αυτές. Ωστόσο, απευθυνθήκαμε και σε μεμονωμένες ε, περιπτώσεις ανθρωπίων δικαιωμάτων. Λάβαμε απαντήσεις, όχι απόλυτα ικανοποιητικέ, αλλά σε μία περίπτωση, εν πάση περιπτώσει, ήταν ικανοποιητική η απάντηση. Σε μία άλλη περίπτωση, όχι τόσο. Αλλά φυσικά είναι μεγάλο θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν θα ήθελα να περιοριστώ στα πολιτικά ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί περιλαμβάνουν φυσικά και τα κοινωνικά και τα οικονομικά ανθρώπινα δικαιώματα. Άρα, να μην περιοριζόμαστε σε συγκεκριμένα άτομα. Είναι θέμα και κοινωνικό. Ασφαλώς και έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά ωστόσο δεν μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, αφού δεν έχουμε το ένα, ας έχουμε το άλλο. Όχι, θέλουμε και οικονομική ανάπτυξη και προσωπικά ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλουμε και τις δύο πλευρές, στο Τουρκμενιστάν και στο παρελθόν στο Ουσμπεκιστάν, εξετάζουν τη δυνατότητα ίδρυσης και άλλων κομμάτων αντιπολίτευσης. Το είπε αυτό και ο Πρωθυπουργό είπε ότι υπάρχει μεν δυνατότητα, αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Στο Τουρκμενιστάν δεν είναι πολύ απλό φυσικά να ιδρύσει κανείς ένα κόμμα αντιπολίτευσης όπως σε άλλες χώρες αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να προωθήσουμε αυτέ τι εξελίξει Και ποια είναι η αντίδρασή του τώρα. ασφαλώ, όπω είπε η Άννα Γκόμες, στο Ουσμπενικιστάν και στο Τουρκμενιστάν συμφωνούμε ότι θα πρέπει να ανοίξει την προσωπία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. να υπάρξει δέσμευση. Κατά δεύτερον, στην ατζέντα έχουμε και την έκθεση Νικολάη, την οποία υπερψήφισε ε, το Κοινοβούλιο. Συμφωνώ ουσιαστικά με όλα όσα αναφέρει. Το ερώτημα όμω που ανακύπτει είναι Πότε. Δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον εισηγητή ακόμα, αλλά πότε θα πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Δύο θέματα θα πρέπει να συνδυαστούν, θεωρώ, και να εξαρτηθούν από αυτά τα ζητήματα η αποδοχή μας ή μη. Το πρώτο εξ αυτών είναι το εξή. Αν θα υπάρξει συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία, από πλευρά Κοινοβουλίου τουλάχιστον θα πρέπει να υπάρχει διάλογο. Ήταν την η πρώτη φορά που συναντηθήκαμε είχε γίνει μία συνάντηση πριν από πέντε χρόνια, αλλά δεν είχαν επιδείξει ενδιαφέρον στην παρουσία μας, για την παρουσία μας. Τώρα υπήρξε κάποιο ενδιαφέρον και ξεκαθαρίσαμε στον Υπουργό Εξωτερικών ότι θέλουμε να υπάρχει και μια ανταπόκριση, ότι θέλουμε να μας επισκεφτούν εδώ στις Βρυξέλλες και μέλη του Κοινοβουλίου στα πλαίσια της συμφωνίας ε, εταιρική σχέσης και συνεργασίας. Και κατά δεύτερον υπάρχει κάποια προθυμία, περιορισμένη ίσως, για την πρόσκληση κάποιων ε, ειδικών απεστελμένων του ΟΗΕ για θέματα παιδείας, βασανιστήριων. Συνεργασία λοιπόν με διεθνείς οργανισμούς. Θα ήταν πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Αν το βάλουμε λοιπόν αυτό στην ατζέντα, σε συνάρτηση με τη Συμφωνία Εταιρική Σχέση. θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στι εβδομάδε πριν αυτή η συμφωνία τα δύο αυτά θέματα. Καταρχάς, η συμμετοχή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων και κατά δεύτερον η συνέχιση των συζητήσεων με τους βουλευτές. Φυσικά ξέρουμε ότι οι βουλευτές στις χώρες αυτές δεν εκλέγονται με τον τρόπο που εκλέγονται σε εμά. Είναι ωστόσο οι συνομιλητές που έχουμε. Αυτά λοιπόν, εν συντομία. Και θεωρώ, το επαναλαμβάνω, ότι είναι απαραίτητη η δέσμευσή μας προς όφελος και της δημοκρατίας, αλλά και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας αυτής, αλλά και προς όφελος δικός μας, δικό μας. Grazie. Ε, il prossimo intervento. Ευχαριστώ. Επόμενη παρέμβαση, η συνάδελφο Κιλ Νίλσεν από του πράσινου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μετά από όσα είπαν οι προλαλήσαντε τα μέλη τη αντιπροσωπείας προηγήθηκαν να μου στο λόγο. Θα ήθελα και εγώ να πω κάποια πράγματα. Η εμπλοκή με το καθεστώς, Φυσικά και δεν μπορεί να γίνει σε βάρο των θεμελιωδών δικαιωμάτων του πληθυσμού. Το είπαν και προλαλήσαντε. Ακριβώ εδώ πρέπει να εμφαθύνουμε και να, να δώσω και εγώ έμφαση σε αυτό. Δεν μπορούμε να δώσουμε εξουσιοδότηση εν λευκό. Το 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση κατήργησε τι κυρώσει που είχε επιβάλει στο Ουσμπεκιστάν μετά την σφαγή του Ντιζάν και θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμή με την ευκαιρία και στα θύματα αλλά και στους ε, εξόριστους μετά την τραγωδία του 2005, γιατί, ε, του Μαΐου του 2009 μάλλον. Γιατί ε, ίσως να έχουν ε, την εντύπωση ότι κλείνουμε τα μάτια ή το στόμα. Εγώ δεν θέλω να κλείσουμε το στόμα και θέλω να το θυμόμαστε αυτό το γεγονός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αποφασίσει το 2009 να υλοποιήσει αυτές τις κυρώσεις, τις περιβόητες κυρώσεις. Κάποιες χώρες, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, είχαν στόχο να επιβληθούν οι κυρώσει αυτές. Τελικά δεν έγινε κάποια διερεύνηση της φαγής αυτής. Δεν υπήρξε επίσκεψη στι φυλακέ. Η καταστολή και η καταπίεση κατά των μέσων ενημέρωση, κατά της κοινωνία των πολιτών, όλο και αυξάνεται. Τελευταίο περιστατικό έκλεισε το γραφείο του Human Rights Watch στην Τασκένδη. Ένα στοιχείο. Ξέρετε ότι το Καζακστάν έχει την προεδρία του 2010, είχε μάλλον την προεδρία του ΑΣΕ το 2010, είχαν δώσει υποσχέσεις για μεταρρυθμίσεις οι χώρες περιοχής. Ξέρουμε όμως τώρα ότι αντίθετα υπάρχει και υποβάθμιση και ε, επιδείνωση των πολιτικών ελευθεριών και αύξηση της καταστολής και της ε, καταπίεσης. Θέλω να τονίσω λοιπόν ότι υπάρχει κίνδυνος να δώσουμε λευκό εξουσιοδότηση σε τέτοιου είδους καθεστώτα. Σημαντική είναι επίσης ε, η χειραγώγηση για την οποία μπορούμε να μας, ε, μάλλον για το, στις οποίες μπορούμε να πέσουμε θύματα. Να σας εξηγήσω, δεν είχα απλά την εντύπωση, ε, κάτι παραπάνω κατάλαβα ότι το ενδιαφέρον που δείχνουμε για την οικολογία και το περιβάλλον ε, ε, οι Ουσμπέκοι δεν ξέρω πώς το κατάλαβαν ακριβώς, αλλά δεν θα έπρεπε να πέσουμε θύματα χειραγώγησης. 15 και το λένε με περηφάνεια ε, έδρες του Κοινοβουλίου είναι για οικολόγους και το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει οικολογικό κίνημα ή κόμμα, ούτε οικολόγια, απλά ε, κάθε περιφέρεια όρισε ποιος θα είναι ο οικολόγος που θα υπηρετεί στο κοινοβούλιο. Για την οικολογία γίνεται πάρα πολύ ε, λόγο. Ε, πράγματι, όπως είπαν συνάδελφοι, το ζήτημα των ε, υδάτων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παραδόξω όμω, το Ουσμπεκιστάν που είναι εντελώ αντίθετο στην περιφερειακή πολιτική, τη δική μα περιφερειακή προσέγγιση και πολιτική, ουσιαστικά απευθύνεται στην Ευρώπη για το θέμα των υδάτων. Μα είπαν ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στα εθνικά σχέδια. Δεν θέλουν περιφερειακή προσέγγιση, θέλουν όμω για τα ύδατα θέλουν να παρέμβουν. Δεν θα πρέπει να μας χειραγωγήσουν γιατί ε, έχουμε κάποια φράγματα, ε, πολύ σημαντικά έργα ε, στο Ραγκούν και γενικώ όλα αυτά τα, έργα και εξοπλισμοί μπορεί να βλάψουν σημαντικά το περιβάλλον. Επίσης, η εντατική καλλιέργεια βαμβακιού στο Ουσμπεκιστάν είναι και αυτός ένας λόγος για το πρόβλημα που υπάρχει με το νερό. Υπάρχει πλήρης επίσης παραγνώριση ε, του συστήματος άρδευσης από πλευρά του Σμπεκιστάν. Δεν θέλω να επεκταθώ, απλά να σας ε, επισημάνω υπάρχει ότι υπάρχει κίνδυνος χειραγώγησης με βάση, ε, μάλλον με άξονα την οικολογία. Ένα άλλο θέμα το οποίο θέλω να αναφέρω για να συμπληρώσω την αναφορά είναι το εξή. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιε χώρε μέλη θεωρούν ότι είναι σημαντικό να έχουν καλέ σχέσει με το Ουσμπεκιστάν και το Τουρκμενιστάν, αυτό το θέλουν γιατί υπάρχει και αυτή η εύκολη πρόσβαση στο Αφγανιστάν, γνωρίζοντας ότι μέσω Πακιστάν από τον Νότο το πέρασμα είναι όλο και πιο δύσκολο και επικίνδυνο. Και πρέπει να το πούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη που έχουν δεσμευτεί σε αυτόν τον πόλεμο στο Αφγανιστάν Μα το λένε ξεκάθαρα, δεν θέλω να κατονομάσω τον πρέσβη, ένα πρέσβη πάντως μα μίλησε για τραυματισμένους στρατιώτες ε, που μπορούν να, επαναπατριστούν από το Αφγανιστάν μέσω του Τουρκμενιστάν. Είναι, το ενδιαφέρει λοιπόν Στη μεθόριο του Ουσμπεκιστάν με το Αφγανιστάν υπάρχει μια αεροπορική βάση, καμιά δεκαριά γερμανικά αεροπλάνα και ελικόπτερα σταθμεύουν εκεί. Υπάρχει μια βάση τέλο πάντων. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη γιατί νομίζω ότι εύκολα ξεχνά κάνει του πραγματικού λόγου για του οποίου εμεί ίσω έχουμε την τάση να είμαστε αρκετά ευνοϊκοί και ευνοϊκά διακείμενοι σε διάφορες σχέσεις, με διάφορα ε, προσχήματα. Αλλά την αλήθεια δεν τη λέμε. Η αλήθεια είναι αυτή το να μπορούμε να εγκαταλείψουμε το κεφάλι ψηλά το Αφγανιστάν. Για μένα είναι δύσκολο, αλλά αυτή είναι η βούληση και βέβαια σε βάρος τελικά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ελευθερίας έκφρασης στην περιοχή αυτή. Αυτό ήθελα να το πω. Και κάτι άλλο σημαντικό. Στις αρχές Μαΐου η κυρία Helen Clark, ε, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του ΠΝΟΥΝΤΑ, επισκέφτηκε και είδε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στη χώρα. Λέει ότι το Τουρκμενιστάν έχει επικοδομητικές εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές. Εγώ διαρωτώ με. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα κατά των βασανιστήριων που εκπονεί μια έκθεση που σύντομα θα δημοσιευθεί και ήδη γνωρίζουμε ότι οι διαπιστώσεις για την πρακτική των βασανιστήριων είναι πραγματικά φρικτές, είναι αποτροπιαστικά τα στοιχεία τα οποία ε, θα λέει η έκθεση. Έχουμε λοιπόν ε, χώρα, μια χώρα όπως το δικάζει που καταδικάζει όλες αυτές τις πρακτικές των βασανιστήριων, αλλά από την άλλη πλευρά να λέγονται κάποια πιο ευνοϊκά λόγια. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη. Και πρέπει να τονίσουμε τις διάφορες αυτές τις πτυχές της συζήτησης. Σας ευχαριστώ. Merci, Κυρία Χάουταλα είναι επόμενη. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα σε αυτά που προείπε η κυρία Γκόμες για το Ουσμπεκιστάν. Με πολύ μεγάλη χαρά συνεργάστηκα και μαζί της και με τον κύριο Σβόποτα και με τους άλλους συναντρέφους στο Τουρκμενιστάν. Αλλά θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο πτυχές ό,τι αφορά το Τουρκμενιστάν. Πρώτα απ' όλα κάποιες παρατηρήσεις για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ήταν κάτι που μας απασχόλησε ιδιαίτερα κύριος Προβέρα θα θυμάται ότι όταν προείδρευε τη συνεδρίαση της Επιτροπής ε, το χειμώνα, ε, είχαμε αποφασίσει να παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυ στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τουρκμενιστάν εν ώψη και της επικύρωσης ε, του PCA. Ίσως να βελτιώνει την κατάσταση, αλλά τουλάχιστον αυτό που παρατήρησα εγώ είναι ότι σχεδόν κανένα θετικό σημάδι δεν υπάρχει, ίσως με την εξαίρεση ότι πιστεύω ότι έχει συνειδητοποιήσει το καθεστώς ότι το να ε, βασίζεται ε, στην, ε, στη βίβλο του πρώην δικτάτορα δεν είναι και κάτι καλό για την οικονομία και την κοινωνία. Άρα υπάρχουν κάποια μηνύματα που δείχνουν ότι ίσως τέτοιου είδους γραφές και ιερά βιβλία θα εξαφανιστούν λίγο-λίγο. Όταν επισκεφθήκαμε το ρωσικό σχολείο, το οποίο με υψηλά δίδακτρα παρακολουθούν παιδιά Ρώσων, εκεί υπήρχε ένα μάθημα που ε, διδάσκονταν τα παιδιά το βιβλίο αυτό του δικτάτορα Νιαζό. Και με εξέπληξε αυτό. Αν όμως δούμε τι έχει υποθεί για την ανάγκη βελτίωση κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εγώ δεν βλέπω να γίνεται κάτι επί της ουσίας. Δεν βλέπω ουσιαστικές αλλαγές. Η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού δεν λειτουργεί ε, με ελευθερία, δεν μπορεί να επισκεφθεί τις φυλακές. Πολιτικοί κρατούμενοι είναι πάρα πολλοί, υπάρχουν περιορισμοί μετακίνησης. Δεν υπάρχει πρόσβαση σε ανεξάρτητους μη κυβερνητικού οργανισμούς, ούτε βέβαια οι φορείς ε, του ΟΗΕ μπορούν να εργαστούν ελεύθερα στη χώρα. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξή. αυτή την κατάσταση, από αυτέ τις περιστάσεις, μήπως θα έπρεπε να ζητήσουμε από του εκπροσώπου μα στο Τουρκμενιστάν αλλά και εδώ στις Βρυξέλλες να ξεκαθαρίσουν ότι πρέπει να δούμε θετικά σημάδια και μετά να επικυρώσουμε τη συμφωνία PCA. Ένα από τα βασικά αιτήματα που έχει ζωτική σημασία κατά την απόψή μου είναι οι ειδικοί εισηγητές των ΗΠΑ να μπορούν να επισκεφθούν τη χώρα και θέλω να τονίσω το ρόλο του ειδικού εισηγητή για τους βασανισμούς. Φαίνεται να υπάρχει ένα πρόβλημα με στα βασανιστήρια που επιμένει στη χώρα και κυρίως στις φυλακές. Το μήνυμα που νομίζω ότι δώσαμε στους πρέσβεϊς των κρατών μελών που επισκεφτήκαμε στο Άσκαμπατ είναι ότι θα πρέπει τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες να σοβαρευτούν πάρα πολύ με ε, τα θέματα των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε επαφέ που έχουν με την κυβέρνηση και το καθεστώς. Έτσι ώστε τελικά να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε κάποια πρόοδο. Δεύτερον, έρχομαι στο θεσμικό ζήτημα. Θα θυμάστε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του στα τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, είχε ζητήσει να υπάρξει ένας ειδικός μηχανισμός παρακολούθησης. Για ποιο λόγο, γιατί πρόκειται για μία από τις πιο καταπιεστικές χώρες στον κόσμο που ασκεί τη μεγαλύτερη καταστολή. Και έχουμε παρόλα αυτά επαφές με αυτή τη χώρα από πολλές πλευρές. Η εξωτερική υπηρεσία, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης δεν δέχθηκε ε, το αίτημά μας να υπάρξει αυτός ο ειδικός μηχανισμός παρακολούθησης. Αυτό έχει ήδη συζητηθεί ήδη στο διευρυμένο Προεδρείο. Ε, πριν από την πράσινη εβδομάδα το συζητήσαμε στο διευρυμένο Προεδρείο της Επιτροπής μας. Και νομίζω ότι μια γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας έχει ζητηθεί. Είναι σημαντική. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η νομική υπηρεσία της ΕΕ θεωρεί ότι ένα ειδικό μηχανισμό παρακολούθησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα στρέβλωνε τη θεσμική ισορροπία. Αγαπητοί συνάδελφοι, Πόσε φορέ τόσα χρόνια έχουμε ξανακούσει ότι ό,τι ζητάει το Κοινοβούλιο στρεβλώνει και διαταράσει τη θεσμική ισορροπία. Σα παρακαλώ να σοβαρευτούμε όλοι. Ποια είναι τα προνόμια μας τελικά. Ποια προνόμια μα έχει δώσει η Συνδίκη τη Λισαβόνας. Το άρθρο 218 κάνει λόγο για τι ε, διεθνεί συμφωνίε Και το Κοινοβούλιο αυτή η διαπραγματευτική εντολή έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν γίνεται κάποια ρητή αναφορά τώρα στο ρόλο των συμφωνιών, άπαξ και εγκριθούν και επικυρωθούν, αλλά νομίζω ότι η διοργανική συμφωνία που έχουμε με, το, με την Επιτροπή θα μπορούσε να δικαιολογεί το να μπορούμε να εκφράσουμε περισσότερες απαιτήσει. Και όχι απλά να πιστεύουμε ότι έτσι θα κάνει τη δουλειά της η ΕΕΔ και θα βελτιώσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πολύ περίεργη είμαι να μάθω αν η νομική υπηρεσία ήδη έχει μελετήσει το θέμα και ποια είναι τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε. Και θα τεθεί προηγούμενο. Είναι η πρώτη συμφωνία εταιρική σχέση και συνεργασία, PCA, που θα εγκρίνουμε με βάση τα προνόμια που μα εκχωρεί η Συνδίκη τη Λισαβόνα και δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε προηγούμενο όπου το Κοινοβούλιο να έχει πολύ λίγε δυνατότητε να παρακολουθεί ότι τηρούνται υποχρεώσει που έχουν αναλυθεί στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν είναι καλό ιονό το ότι ε, τα ορόσημα τα οποία έχουμε πολλέ αναφέρει, τα σημεία αναφορά ε, που έχουμε αναφέρει πολλέ φορέ για το Τουρκμενιστάν, δεν τα τηρεί η χώρα. Παρ' όλα αυτά η ΕΕΔ θεωρεί ότι πρέπει να επικυρώσουμε αυτή την ε, συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, PCA. Νομίζω ότι πρέπει και εμείς να φροντίσουμε τα δικά μας θεσμικά συμφέροντα και δικαιώματα για να βελτιωθεί η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μία από τις χώρες όπου βλέπουμε τη μεγαλύτερη καταστολή. Ευχαριστώ. επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Γέγκλε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους καταρχήν, την κυρία Γκόμες και τον κύριο Σβόμποντα ε, για την ε, αναφορά που μας έκαναν για τις επισκέψεις αυτές στο Σμπεκιστάν και στο Τουρκμενιστάν. Είμαι μέλος της αντιπροσωπείας από το 1999, της αντιπροσωπείας για την Κεντρική Ασία. Και έκτοτε έχω διαπιστώσει ότι έχουν υπάρξει πρόοδοι, οπισθοχωρήσεις, αλλά και νεκρές περίοδοι. Όσον αφορά το Ουσβεκιστάν, θα ήθελα να πω ότι όλα ένα και περισσότερο η στάση μου είναι πιο θετική. Γιατί, ναι, είναι πολύ δύσκολη η χώρα αυτή. Ε, είναι όμως δυνατόν να ξαναρχίσει η συζήτηση και η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού μπόρεσε να μπει στις φυλακές εδώ και κάποια χρόνια. Το Ουσμπεκιστάν έχει καταργήσει τη θανατική ποινή και έχει δημιουργήσει στην νομοθεσία του κάποιες διατάξεις που εμείς ζητήσαμε. Φυσικά θα χρειαστεί να περιμένουμε κάποιο διάστημα πριν να εφαρμοστεί πλήρως η νομοθεσία αυτή και πριν να ενσωματωθεί και η νοοτροπία θα πρέπει μάλλον να περιμένουμε ακόμα μια γενεά πριν να τα καταφέρουμε. Είναι πολύ σημαντική η πρόκληση λοιπόν στον τομέα αυτό. Κάτι ακόμα σημαντικό είναι ότι όλες οι χώρες της Κεντρικής Ασίας, όλες θα πρέπει να κληθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους όσον αφορά την ενέργεια και την, ε, τον ανεφοδιασμό σε νερό. Πρέπει από κοινού να διαχειριστούν το πρόβλημα αυτό. Επιπλέον μια χώρα όπως το Ουσμπεκιστάν οφείλει να μεριμνήσει ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί τα εσωτερικά του προβλήματα όσον αφορά την, τον ανεφοδιασμό νερού. έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των παλαιών ε, καναλιών ε, της ε, πρώην Σοβιετικής Ένωσης, όπου υπάρχουν τρομερές διαρροές και χάνεται πολύ νερό. Το Καζαστάν ήταν υπεύθυνο για τις πρώτες ύλες της Σοβιετικής Ένωσης. Το Ουσβεκιστάν ήταν υπεύθυνο για τα, τις ζωοτροφές και τη θέρμανση. Έτσι τα έχει οργανώσει η Σοβιετική Ένωση. Όμως σήμερα η κατάσταση φυσικά δεν είναι πλέον η ίδια. Υπάρχει ε, διαφοροποίηση ανάμεσα στις διάφορες χώρες ε, που ε, περιπλέκει τα πράγματα. Μετά από το σεισμό στην Ιαπωνία θα πρέπει να διαρωτηθούμε αν και κατά πόσο μια τέτοια υποδομή τόσο ογκώδης είναι καλή τελικά. Και η Παγκόσμια Τράπεζα εξετάζει το θέμα και σίγουρα θα μας δώσει κάποιες πληροφορίες για το θέμα αυτό. Θα πρέπει να λάβουμε πολύ στα σοβαρά τη στρατηγική μας στην Ασία και θα πρέπει να συμφωνήσουμε για τις προτεραιότητές μας. Αυτό για όλες τις χώρες σημαίνει οικονομική ανάπτυξη κοινωνική ανάπτυξη και το είπε με σαφή τρόπο ο κ. ότι από αυτό εξαρτάται και ο εκδημοκρατισμός και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό ισχύει για όλους, σε διαφορετικό βαθμό, αλλά αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να πατήσουμε από όλους. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, ούτε θα πρέπει να κάνουμε εξαιρέσεις, ούτε για το Τουρκμενιστάν. Όντως, η πρώτη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ε, ε, είναι τώρα, μετά τη Λισαβόνα. Δεν είχαμε πριν τέτοιες δυνατότητες. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχουμε καλύτερες δυνατότητες να απαιτήσουμε συγκεκριμένα στοιχεία χωρίς συμφωνία εταιρικής σχέση, σχέσης. Δεν έχουμε πραγματική δυνατότητα να συνεισφέρουμε. Οι απαιτήσει που θέτουμε προκειμένου οι κυβερνοβουλευτικές επιτροπέ να έχουν τακτική λειτουργία είναι κάτι το αυτονόητο. Και αυτό θα πρέπει να το πετύχουν οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου μας. Και θα πρέπει να πετύχουμε να είναι δυνατή η επίσκεψη από μέλη του Κοινοβουλίου του Τουρκμανιστά. Όπως και για παράδειγμα η ανταλλαγή και οι επισκέψεις από ε, νεαρά άτομα όπως γίνεται και σε άλλες χώρες, προκειμένου να εξάγουμε, αν θέλετε, τη γνώση μας. Και θεωρώ ότι αφενός θα πρέπει να απαιτήσουμε και να υποστηρίξουμε με έξυπνο τρόπο τις χώρες εκείνες. Αν το καταφέρουμε αυτό, θα λάβουμε κι εμείς κάτι ως ε, αντίκρισμα. Και ομολογώ ότι είμαι Γερμανίδα και ότι δεν απέχω πάρα πολύ και ότι έχω ευθύνη σε ό,τι αφορά το Ουσμπεκιστάν, σε ό,τι αφορά τους Γερμανούς στρατιώτες για τις οικογένειές τους. Και που και που πηγαίνουν και σε κηδείες. Και αυτά δεν είναι απλά πράγματα. Και εδώ απαιτείται ένα πνεύμα κοινό και όχι απομόνωσης. Αυτό το απευθύνω σε έκκληση στην Επιτροπή μας. Τελευταία παρέμβαση της συνάδελφος Νικολάη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως εισηγήτρια συμμετείχα στην επίσκεψη στο Τουρκμενιστάν στην αντιπροσωπεία της οποίας ηγήθηκε ο κύριος Βόμποντα και ήθελα να τον ευχαριστήσω για τον τρόπο με τον οποίο ηγήθηκε της αντιπροσωπείας. Ήθελα να, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και για όσους παρακολούθησαν πρώτη φορά ε, τέτοια αντιπροσωπεία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Ο κύριος Βόμποντα θύμισε το γεγονός ότι θα ήθελε να έχει περισσότερα κόμματα αλλά ότι ο κόσμος δεν το επιθυμεί. Εγώ προέρχομαι από μια παλιά κομμουνιστική χώρα και, έλεγα, και θυμάμαι ότι ο δικτάτορας Τσαουσέσκου έλεγε αυτό το πράγμα, ότι δηλαδή ο, εκείνος ήθελε περισσότερα κόμματα αλλά ο κόσμος δεν το ήθελε. Ε, ας μην το ξεχνάμε αυτό πρέπει να συγχαίουμε τα πολιτικά καθεστώτα με τα έθνη και με τους λαούς. Μπορούμε να καταδικάζουμε το καθεστώς και φυσικά το καθεστώς του Τουρκμενιστάν είναι τελείως κατακριτέο ακόμα κι αν το προσπαθεί να κάνει πρόοδο προς δημοκρατικά στάνταρ και προδιαγραφές αλλά είναι βέβαιο ότι μπορούμε να ασκήσουμε πολλές επικρίσεις. Δεν μπορούμε ωστόσο να να, καταδικάσουμε το λαό μόνο και μόνο επειδή έχει τέτοιο καθεστώς. Πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία στο λαό αυτό. Ε, να εξάγουμε αν μπορέσουμε το πρότυπο δημοκρατίας γιατί η έλλειψη αποφασιστικότητας δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να έχουν άλλη επιλογή. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι παρούσα επιτόπου μέσω μιας ε, ε, διπλωματικής αντιπροσωπείας το 20 ε, της Ευρώπης κάνει κάποια πράγματα τα Ηνωμένα Έθνη επίσης και μπορέσαμε μάλιστα να δούμε τα προγράμματα του ΟΗΕ και τα αποτελέσματα αυτών των προγραμμάτων που είναι πολύ εθαρρυντικά. Αλλά η παρουσία μας εκεί είναι απαραίτητη για να στηρίξουμε ακριβώς τον λαό αυτό. Πρέπει να δείξουμε σε αυτό το λαό το δρόμο γιατί εάν δεν το γνωρίζει δεν μπορεί να διακρίνει ένα πρότυπο δημοκρατίας. Δεν μπορούμε να ζητάμε από τον λαό να έχει υψηλέ προσδοκίες άμα δεν, γνωρίζει, δεν γνωρίζει καν το πρότυπο λόγω του μπλοκαρίσματος, ε, λόγω της παρεμπόδισης της ενημέρωσης ε, ε, που γίνεται από αυτό το καθεστώς. Αυτή η εμπειρία, η εμπειρία που έχουμε εμείς από κομμουνιστικές χώρες την ξαναβρίσκουμε σε αυτές τις χώρες. Το Τουρκμενιστάν είναι η μόνη χώρα η οποία δεν, δεν έχει υπογράψει συμφωνία συνεργασίας. Η κυρία Γκόμες μίλησε και για το Ουσβεκιστάν που επίσης έχει προβλήματα, αλλά τουλάχιστον επωφελείται από μια ε, συμφωνία συνεργασίας. Η χώρα αυτή λοιπόν πρέπει να συνδεθεί με τα ευρωπαϊκά στάνταρ και πρέπει να τη στηρίξουμε. Πιστεύω πως μέσω τροπολογιών μπορούμε να θέσουμε όρους και τουλάχιστον σε αυτή την φάση δεν αμφιβάλλω για την ε, ικανότητα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης να θέσει σε εφαρμογή κάποιους κανόνες για μια τέτοια συμφωνία. Πιστεύω ότι οφείλουμε να επανεπικυρώσουμε την εντολή αξιοπιστίας και εμπιστοσύνη που έχουμε δώσει σε αυτή την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, να επαναλάβουμε την εμπιστοσύνη μας και επίσης κάνω έκκληση για ένα άνοιγμα από πλευράς μας προς ένα μελλοντικό νομικό πλαίσιο γιατί είναι ο μόνος τρόπος να είμαστε αποτελεσματικοί στις δράσεις μας σε αυτές τις χώρες. Ε, το κοινοβουλευτικό άνοιγμα και το διπλωματικό άνοιγμα θα πρέπει να είναι μια λύση για αυτές τις χώρες. Είναι μια από τις πιο σημαντικές αντιπροσωπείες αυτή που μετέβει τώρα στο Αξαμπάτ και ε, πραγματικά θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τις ιδέες μας και τις αρχές μας επί τόπου. Οι αρχές του Τουρκμενιστάν ήταν αρκετά ανοιχτέ, ακόμα και αν μας παρουσίασαν την κατάσταση με αρκετά τυπικό τρόπο, σοσιαλιστικό τρόπο ε, και φυσικά μας είπαν ναι, ξέρουμε ότι απέχουμε από τα δημοκρατικά στάνταρ αλλά πρέπει να τους στηρίξουμε στην πορεία τους γιατί διαφορετικά αν μείνουμε εκτός αν δεν εμπλακούμε θα διατηρηθεί το status quo, πράγμα το οποίο δεν είναι προς το συμφέρον αυτού του λαού και ούτε και προς το δικό μας συμφέρον φυσικά. Νομίζω λοιπόν πως μπορούμε να συζητήσουμε μια ολόκληρη σειρά τροπολογιών ώστε η διαδικασία αυτή να καταστεί πιο αποτελεσματική και να ξεκινήσουμε μια διπλωματία καλής πίστης ώστε αν θέλουμε να είμαστε ορατοί και αποτελεσματικοί, να μπορούμε να είμαστε παρόντες επί τόπου. Διαφορετικά οι όσοι έχουν άλλα πρότυπα να προτείνουν, όπως η Ρωσία και η Κίνα, που βρίσκονται στην περιοχή, ούτως ή άλλως θα εξάγουν τα δικά τους πρότυπα και θα έχουμε χάσει έτσι την Κεντρική Ασία. Έχουμε λοιπόν μια ευθύνη ως ε, κράτη τα οποία θέλουν να εξάγουν ένα δημοκρατικό πρότυπο σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μια σύντομη παρέμβαση από την συνάδελφο Γκόμας. Παρακαλώ. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που μίλησαν για το Ουσμπεκιστάν. Δεν θα ήθελα όμως να επανέλθω στο Τουρκμενιστάν. Με εντυπωσίασε το δάσος δορυφορικών ε, πιάτων πάνω στα κτίρια. Παρά το γεγονός ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι και απαγορευμένοι, δεν επιτρέπονται. Αυτό νομίζω ότι υποδεικνύει ότι ο κόσμος έχει κάποια εκπαίδευση, εν πάση περιπτώσει ενημερώνεται για το τι συμβαίνει. Και αυτό μου έκανε εντύπωση. Η αξιωματούχοι φαίνεται ότι είναι όμοιροι των ατόμων εκείνων που τους παρακολουθούν, από ό,τι φαίνεται. Πιστεύω φυσικά ότι και στο Ουσμπεκιστάν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει και κάποιος βαθμός εκλεπτισμού, αν θέλετε, για τα πράγματα εκείνα που ακόμα δεν έχουν επιτευχθεί στο Τουρκμενιστάν. Νομίζω ότι η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης δεν θα αλλάξει τη δέσμευση που χρειαζόμαστε. Συμφωνώ και εγώ με τους συναδέλφους ότι τη χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε δέσμευση, χρειαζόμαστε μια σωστή αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπε ο κ. Σβόποντα, αλλά η συμφωνία εταιρική σχέσης θα νομιμοποιούσε κατά τρόπον ε, την κυβέρνηση αυτή, κατά τρόπο που δεν αξίζει ενδεχομένως, γιατί δεν έχουμε πετύχει τα ορόσημα που θέλουμε και μου έκανε εντύπωση και πάλι να τονίσω ότι χρειαζόμαστε μια αντιπροσωπεία με αξιωματούχους οι οποίοι θα είναι υπόλογοι σε εμάς, όχι με άτομα που θα φοβούνται για τη δουλειά τους. Που δεν θα τολμούν τις ερωτήσεις που πρέπει. Ιδάλλως δεν θα υπάρχει καμία αποτελεσματικότητα. Άρα, θα υποστηρίξω τα σχόλια του κυρίου Σβόμποντα, ότι δεν θα πρέπει να βιαστούμε σε καμία περίπτωση για να υπογράψουμε τη συμφωνία αυτή. Ο... Συνάδελφος Σβόμποντα, χωρίς να ξαναρχίσουμε τη συζήτηση. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Μία μικρή υπότεξη να κάνω. Όλε οι γειτονικέ χώρες είναι μη δημοκρατικέ του Τουρκμενιστάν. Τέσσερι ενδεχόμενοι εταίροι η ΙΠΑ, οι οποίες τελικά το μόνο που τις ενδιαφέρει είναι η πρόσβαση στο Αφγανιστάν. Η Κίνα είναι μια χώρα η οποία δεν δεσμεύεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ρωσία το ίδιο. Ο μοναδικός εταίρος ο οποίος κάτι θα μπορούσε να κάνει για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι η Ευρώπη. Ας είμαστε ειλικρινείς. Ας προσπαθήσουμε να πετύχουμε τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας με κάποια στοιχεία, γιατί είμαστε οι μοναδικοί εταίροι οι οποίοι θα διαφερθούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, να σα θυμίσω ότι την 5η 26 θα γίνει μια ακρόαση τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για τη Στρατηγική στην Κεντρική Ασία. 5η 26. Από τις 9 μέχρι τις 11 προβλέπεται αυτή η ακρόαση. Τώρα, πριν την ψηφοφορία... Come?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 Colleghi. Quando dobbiamo saltare ti dico eventualmente qual è sì. il prossimo. Così. Abbiamo le votazioni elettroniche. Su... Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για κάποιες εκθέσεις. Λοιπόν, ξεκινάμε. με την πρώτη έκθεση κύριου Βανόρντεν. Παράγραφος 2, συμβαστική τροπολογία παριθμών 6, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά ή μάλλον υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική υπερθμόν 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41 τώρα. Παρακαλώ. Μα ε, κάτι δεν έχω καταλάβει. Τι έγιναν με τις συμβιβαστικές 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7. Έρχονται αργότερα. Στον κατάλογο ψηφοφορίας ε, έχουμε μια διαφορετική σειρά. Έχουμε ε, εντελώς διαφορετική με αρρύθμιση. Μα πού είμαστε κύριε Πρόεδρε, δεν έχω χαμένα, τα έχω τελείως χαμένα. Κύριε Πρόεδρε, για εμάς που μόλις φτάσαμε, ε, θα ήθελα να μας πείτε πού βρισκόμαστε. Επειδή είμαι συγγετής, όπως καταλαβαίνετε, ενδιαφέρομαι όλος ιδιαίτερος να ξέρω σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Λοιπόν, πού είμαστε. Είμαστε στην πρώτη σελίδα του voting list. Πράγματι, τη δική σας έκθεση ψηφίζουμε, κύριε Φανόρτεν, και είμαστε στην τροπολογία 41. Μα τι έγινε με τις συμβιβαστικέ. Οι 6 και 7 έχουν εγκριθεί. Yeah, yeah, they, και Μα ο κατάλογος ψηφοφορίας, το voting list που έχουμε εμείς είναι τελείως διαφορετικό. Λοιπόν, τροπολογία 41. Και 41. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 τροπολογία υπέρ κατά. Ε, πρέπει να το ελέγξουμε. Για την τροπολογία 42 ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται και αυτή. 45 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά τη 45. Λοιπόν, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 45. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 49. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά. Ελεκτρονικά παρακαλώ. την 50. Την τροπολογία 50 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Και αν κάποιο θέλει να ψηφίσει προφορικά μπορεί να το κάνει. Λοιπόν, 9 συμβιβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 55 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 58 τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Ας το ελέγξουμε. Ας το ελέγξουμε. Τροπολογία 61. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με 36 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 62 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 63 τροπολογία υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 64 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11 Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 67. 67. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 68, όχι 70. Ποιοι είναι υπέρ της 70. Κατά. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να ελέγξουμε την 70, άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με μία μόνη εις ψήφο διαφορά. Δεν είχα την κάρτα μου, λέει η κυρία Λάτφορντ. Αν είχα την κάρτα μου θα είχα ψηφίσει υπέρ. Βέβαια πάλι θα είχε απορρίφθει, αλλά τέλος πάντων. Γιατί θα είχαμε ισοψηφία. 27 όλα. Λοιπόν, συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 75 υπέρ. Κατά. Ε, ε, γίνεται δεκτή. Τώρα τι ψηφίζουμε. Θέλετε να το ελέγξουμε, ας το ελέγξουμε. Την 75 αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 80. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 81 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Θα ελέγξουμε. Ηλεκτρονικό έλεγχο για την τροπολογία 82. Chiusa la votazione. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 83. Και a 83. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 84 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 85 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 86 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 87 Α, για την 86 ελέγχουμε, ηλεκτρονική ψηφοφορία, Votazione elettronica chiusa. Τέλος ψηφοφορίας. Πρέπει να προσθέσουμε μία ψήφο κατά, αλλά εγκρίνεται. 87 in parte 87 χωριστά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά. Ελέγχουμε. Ελεκτρονικός έλεγχος για το πρώτο τμήμα της 87. Elettronica chiusa. È approvato di un voto. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Δεύτερο τμήμα της 87 υπέρ. Και contrario. Respinto. Κατά. Απορρίπτεται. 88. 88. Συγγνώμη, διορθώνει ο πρόεδρος. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 88 υπέρ. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 88, γιατί δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ελέγχω, ελέγχω. Απέρτα la votazione elettronica. Chiusa la votazione elettronica. Τέλος της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 89 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 90 έχει αποσυρθεί. Η 91 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 92 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 15. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 16. Όχι, η, τρι, η συμβαστική 3. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά απορρίπτεται. 20 όχι, 22 με συγχωρείτε, 22 Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 19 ζητήθηκε. Ψηφίζουμε. Avete votato, la votazione è chiusa. Ψηφίσατε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Passiamo al 22. Passiamo al 22. 22 τώρα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά εγκρίνεται 24 υπέρ κατά εγκρίνεται 25 υπέρ κατά απορρίπτεται 26 υπέρ κατά εγκρίνεται 27 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 27. Τέλος πληροφορίας. Απορρίπτεται. Έχουμε ισοψηφία, οπότε απορρίπτεται. 28. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Εντάξει, ας ελέγξουμε. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εντάξει, ένα ορεκτικό. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Εδώ έχουμε αμφιβολία. Λοιπόν, ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 1. Λείπει μία ψήφος. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. Στη 2 τώρα. Υπέρ. Κατά. Μα σηκώντε τα χέρια σας γιατί διαφορετικά δεν καταλαβαίνω. Τροπολογία 2. Παρακαλώ σηκώστε τα χέρια όσοι είστε υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται με πλειοψηφία. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. κατά εγκρίνεται. Περνάμε συμβαστική 1, ποιοι είναι υπέρ, κατά εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. Ε, με ηλεκτρονική ψηφοφορία θα ψηφίσουμε. Σας παρακαλώ να ψηφίσετε τώρα. Τέλος της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Παρακαλώ, ο κύριος Φανόρδεν. Καταρχήν, Πρόεδρε, να εκφράσω την ε, ευγνωμοσύνη μου στα μέλη για την υποστήριξή του. Θα ήθελα απλώ να καταγραφεί η ανησυχία μου για τον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτή η ψηφοφορία. Διότι ο κατάλογο ψηφοφορία που είχαμε είναι διαφορετικός από αυτόν με βάση τον οποίο εργαστήκαμε μέχρι το μεσημέρι σήμερα. Δεν ξέρω τώρα πώς έγινε αυτό, αλλά με ανησυχεί για, ως εισηγητής να καταλήγουμε σε έναν κατάλογο ψηφοφορίας όπου δεν αναγνωρίζουμε τίποτα και όπου έχουν ανακατευτεί παράξενα όλα αυτά. Ποιος το, ε, ποιος το εφήβρε, πώς ε, φτάσαμε σε αυτό. Μπορείτε να μου πείτε πότε λοιπόν ξανασυστάθηκε αυτό ο κατάλογο ψηφοφορία με αυτή τη σειρά. Διαβίβασα την ανησυχία σα στη γραμματεία και θα σα δώσουμε περιστατωμένη απάντηση Μόλι θα έχουν δει ακριβώ τι συνέβη. Θα σας απαντήσουν συντόμως. Να σας πω εγώ τώρα, εγώ ίδιος δεν ξέρω τι συνέβη. Λυπούμε. Um, ναι, να πω και εγώ δύο λόγια, Πρόεδρε. Πριν αρχίσετε με την επόμενη ψηφοφορία, να σας πω τα εξής. Καταρχήν, θέλω να έχω το λόγο στο τέλος για την προφορική τροπολογία μόνο 1. Εκεί όπου προτείνεται μια αλλαγή και ενώ έχω το λόγο δεν είμαι και τόσο εξοργισμένη αλλά να εκφράσω μια κάποια απογοήτευση, γιατί έπρεπε να καταψηφίσουμε τέσσερις από τις υποτιθέμενες συμβιβαστικές τροπολογίες για αυτή τη γνωμοδότηση, γιατί κατά τη γνώμη μου δεν ήταν πραγματικά συμβιβαστικές και οι τροπολογίες τις οποίες υποτίθεται ότι συμπεριλάμβαναν ή απορροφούσαν, δεν έχουν πραγματικά αντικατοπριστεί σε αυτές τις υποτιθέμενες συμβιβαστικές. Λυπούμε γι' αυτό. Δεν θυμάμαι καμιά έκθεση που να έχει κάνει η Άλντε, ε, όπου θα χρειαστεί να καταψηφίσουμε το 80% των συμβαστικών τροπολογιών, αλλά φοβούμαι πως αυτό θα κάνουμε. Θέλω να απαντήσω σε αυτό, Πρόεδρε, άμα επιτρέπετε. κοιτάξτε, συγγνώμη συνάδελφε, πρώτα ζήτησε να παρέμβει ο συνάδελφος Βιγγένεν, στον οποίο... Βιγγενίν, στον οποίο θα δώσω το λόγο και μετά θα πάρετε και εσείς το λόγο. Να απαντήσω στον κύριο Φανόρντεν ότι ο κατάλογος ψηφοφορίας ήταν ανέκαθανα έτσι. Πόσο ο κύριος Βαν πήρε άλλο κατάλογο. Μήπως ψηφίσατε για διαφορετική έκθεση. Για μας είναι έκπληξη το ότι έχετε κάτι διαφορετικό μπροστά σας. Θα περιμένω από τη γραμματεία να μου απαντήσει για το πότε έγινε αυτή η αλλαγή στη κατάλογο ψηφοφορία. Σίγουρα εμείς δεν δουλεύαμε πάνω σε αυτόν. Και για να απαντήσω στο όσα είπε η Σάρα Λάτφορντ, Νομίζω ότι οι σκιώδεις ηγητές ε, θα συμφωνήσουν ότι κάναμε διάφορες συνεδριάσεις ε, για την έκθεση αυτή και συζητήσαμε τις συμβιβαστικές. Α, ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Εντάξει, το αποσύρω αυτό. Ο συνάδελφος Μποτικόφερ. Μία μικρή ασάφεια, Πρόεδρε. Υπήρξε μία μικρή ασάφεια γιατί στον κατάλογο ψηφοφορία, για παράδειγμα στην τροπολογία 1, έχουμε την σύσταση του κυρίου Φανόρντεν ε, θετική. Και ο βουλευτής Φανόρντεν ζήτησε να την καταψηφίσουμε τελικά την ε, τροπολογία, άρα να τις διευκρινίσουμε αυτές τις ασάφειες. Eh, Εγώ θέλω να σας ζητήσω να διακόψουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων, γιατί διαφορετικά δεν θα φτάσουμε στο τέλος της ψηφοφορίας. Επιπλέον πιστεύω ότι ο κατάλογος ψηφοφορίας δόθηκε αρκετά έγκαιρα. Δεν είχαμε καμιά αμφισβήτηση η ε, ούτε παράπονα ακούσαμε πριν από την ψηφοφορία και γι' αυτό και ξεκίνησα την ώρα που είχαμε προβλέψει την έκθεση με βάση τον κατάλογο ψηφοφορία που έχω στα χέρια μου και που εσείς έχετε στα χέρια σας. Θα έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις ψηφοφορίες μας και έπειτα αν υπάρχουν ε, κάποιες ε, διαμαρτυρίες φυσικά και θα τις σημειώσουμε. Allora, il, passiamo Περνάμε τώρα στην ε, ψηφοφορία για την έκθεση Hankins. Η αντιτρομοκρατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βασικά επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Δύο λείπουν από την ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Κατά. Εγκρίνεται. Επτά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 13 ε, υπέρ κατά απορρίπτεται. Ε, εντάξει, θα ζητάω, θα ρωτάω κιόλα ποιοι απέχουν τις αποχές. Αποχές. Εντάξει, το σημειώνουμε. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Επέρα. Ε, ε, I'm very sorry. Λυπάμαι. Ναι, καταγράφουμε τη ψήφο σας. Κοιτάξτε. Ο κανονισμός προβλέπει ότι από τη στιγμή που έχουμε ολοκληρώσει την ψηφοφορία και αφού έχουν καταγραφεί και οι ψήφοι, δεν μπορούν να, γίνουν, να, δοθούν δεύτερες ευκαιρίες. Αυτός είναι ο κανονισμός που ισχύει νομίζω και σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια και γι' αυτό αυτό τον κανόνα θα ακολουθήσω. Τροπολογία 15. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17. Υπέρ. Τι να κάνουμε, πάμε πίσω στη 15. Στη 15. 15, εντάξει. Ας πάμε πιο αργά. από εδώ και μπρος θα πηγαίνουμε λίγο πιο αργά. Τροπολογία 15, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Allora... Sì, chiudo la votazione. Ναι, τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Emendamento 17. Τροπολογία 17. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Δεκαοχτώ έχει αποσυρθεί. Quindi emendamento orale 2. Προφορική τροπολογία υπαριθμών 2. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ αποχές ποιος είναι κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 28 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιο είναι υπέρ,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 κατά αποχές εγκρίνεται 35 δεύτερο τμήμα ποιο είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 39. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τρο... Συμβαστική 5. Υπέρ κατά Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Συμβαστική 5. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λείπει μία ψήφος. Εντάξει. Τέλος ψηφοφορίας. Είναι σαφές ότι εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. Τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το λόγο έχει για την προφορική τροπολογία η συνάδελφος Λάτφορντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η προτινόμενη προφορική τροπολογία θα ήθελα να ψηφιστεί μόνον εφέσεων έχει τις λέξεις ε, σε έντονους χαρακτήρα, ότι δηλαδή επισημαίνει την ανάγκη να υπάρξουν συμφωνίες κατά τη τρομοκρατία με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον υπάρχει σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να προσθεθούν δηλαδή οι λέξεις με έντονους χαρακτήρες η εισηγήτρια δεν είναι εδώ, ε, μέρους της. Θα ήθελα να πω το εξής. Ξαναδιάβασα πάρα πολύ προσεκτικά και συγκεκριμένα Μιλάμε για strategic partnerships, στρατηγικές εταιρικές σχέσεις εκτός Ευρώπης. Αν μιλάμε για αυτό, καλό είναι να απαιτηθεί ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν μιλάμε όμως απλά για ανταλλαγή πληροφοριών. Όχι, αλλά αν μιλάμε για κάτι τόσο γενικό, συνολικό, νομίζω ότι η ομάδα μου μπορεί να στηρίξει την προσθήκη αυτή. Στρατηγική εταιρική σχέση με την Κίνα είναι ένα παράδειγμα. Βέβαια, εκεί ίσως να έχουμε προβλήματα. Άρα καλό να το προσθέσουμε. Ή με το Ιράν, σωστά. Άλλο ένα καλό παράδειγμα θα μπορούσαμε να δεχθούμε ίσως το occasional information. Ενίοτε να υπάρχει ενημέρωση, πληροφόρηση. Λοιπόν, το στηρίζουμε αυτό που είπε η κυρία Λάτφορντ. Ωραία, ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία που προτείνει η συνάδελφος Λάτφορτ, όπως μας το εξήγησε και το, ανέδειξε, ε, το υπέδειξε μας. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά το σύνολο της ε, γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Okay. Μάνκανο Λοιπόν, τρεις συνάδελφοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με μεγάλη πλειοψηφία. Bene, allora passiamo alle successive. Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Η συγγήτρια είναι η κυρία Μουνής Δεορκίσα. Είναι η εντολή για το τριμερή διάλογο. Έχετε τον κατάλογο ψηφοφορία ενώπιον σα. Ε, ξεκινάμε με την τροπολογία 1 τη συναδέλφου Λόζινγκ Περ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία, ε, συγγνώμη, 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 της συναδέλφου Γκόμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Αποχές κατά. 16 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ε, ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 17 ψηφίζουμε. ΟΚ. votazione chiusa. E Τέλος της ψηφοφορίας απορρίπτεται συμβεβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Emendamento 23. Chi è Τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 26 άρχεται η ψηφοφορία τέλος της ψηφοφορίας ε, απορρίπτεται 27 υπέρ Κατά. Αποχές έγκρινεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Τελική ψηφοφορία. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. 56 ε, υπέρ 1 κατά 6 αποχές. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Τελευταία ψηφοφορία. Ε, ε, Εδώ η συγκεκριτής είναι ο κύριος Μπροκ. Παρα... Τροπολογία 4, παράγραφος 1, υπέρ. Κατά απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στο 5. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 5 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στη 13. Προφορική τροπολογία. Ποια είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 15. Όχι. Συμβιβαστική 2. Με συγχωρείτε. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Πάμε στην 24. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26. Χωριστή ψηφοφορία εδώ, κατά τμήματα δηλαδή, ε, ψηφίζουμε για το πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 ε, κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 39. Όχι, πάμε στην συμβαστική 7, γιατί τη συμβαστική 1 την υιοθετήσαμε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη 42. Τροπολογία 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία... Μάλλον, συμβιβαστική 9. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονική ψηφοφορία. Δεν βλέπω πολλά χέρια ψηλά για τη συμβαστική εννέα. Ποιοι είναι υπέρ και ποιοι είναι κατά. Για πείτε μας ηλεκτρονικά. Λοιπόν, δύο συνάδελφοι, ένας, τέλος ψηφοφορίας. Έγκρινεται με μεγάλη πλειοψηφία. Και περνάμε στην τροπολογία 46 ε, ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Εντάξει. Ηλεκτρονική ψηφοφορία αφού το ζητάτε. Δεύτερο τμήμα της ε, τροπολογίας 46. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 50 όχι λάθος περνάμε συμβαστική 10 συμβαστική 10 υπέρ ποιοι είναι κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 57 με χωρίς τη ψηφοφορία πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 Δεύτερο τμήμα της 57 ζητήθηκε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Manca un Λείπει ένα συνάδελφο. Τέλο ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε στη 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα αν μπλοκ της 1, 2, 3. Υπέρ. όχι, δεν συμφωνούνε. Δεν συμφωνείτε. Ποιος είναι κατά. Όχι. Λοιπόν, χωριστά τις τροπολογίες. Υπέρ. Ποια είναι υπέρ του 1. Ε, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροποποιημένη πρόταση. Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 58 υπέρ 3 κατά. Καμία αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν με μεγάλη πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Colleghi, passiamo al punto 9. In congiunta con la... Σημείο 9, συνάδελφοι. Αποκινούμε την Υποεπιτροπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σημείο 9. Εξωτερικέ πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ του εκδημοκρατισμού. Vorrei informare i colleghi να ενημερώσω τους συναδέλφους το σημείο 9 αναφέρεται στην πρώτη εξέταση στην Επιτροπή Εξωτερικών της έκθεσης για τις εξωτερικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ του εκδημοκρατισμού. Είναι μια έκθεση την οποία ε, συντάσσει η κυρία Βερονίκ Ντεκεζέρα. Έχουν υποβληθεί 235 τροπολογίες στο σχέδιο έκθεσης. Έχουν ήδη γίνει δύο συζητήσεις, μία στην Επιτροπή Δικαιοσύνης και μία επί τη βάση της, ε, του, του, εγγράφου εργασίας και μία άλλη επί τη βάση της έκθεσης να δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειές μας για το μέλλον είναι ο στόχος και πριν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Τικεζέρ, θα ήθελα να θυμίσω ότι αν χρειαστεί η συζήτηση περί τροπολογιών θα συνεχιστεί στην για το τέλος της συνεδρίασης στις 26 Μαΐου και η συνεδρίαση, μάλλον η ψηφοφορία, προβλέπεται στο Στρασβούργο στις, 20, ε, στις 2 Ιουνίου και στην Ολομέλεια θα περάσει από την Ολομέλεια του Ιουλίου. Παρακαλώ, θέλετε κάτι να πείτε για την ημερήσια διάταξη. Σας παρακαλώ. Allora, la parola al relatore. Το λόγο έχει η συγγήτρια λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είχα ήδη την ε, ευκαιρία να σας εκθέσω το στόχο και τη δομή της έκθεσης. αλλά και τη σημασία που έχει στο πλαίσιο το πολιτικό το υφιστάμενο. Άρα να μην επανέλθω σε αυτά. Απλά θα ήθελα να σας μιλήσω για την συνεργασία με τους κοινότητες συζητητές και ακριβώς για αυτές τις 237 τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές που στις πολιτικές τους ομάδες ε, κατέθεσαν μια σειρά τροπολογιών, ο καθένας, η καθεμία που θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, χωρίς να ε, καμία αυταρέσκεια, που συμβάλλουν πραγματικά στη βελτίωση, τη σημαντική βελτίωση της έκθεσης. Υπάρχουν κάποιες αποχρώσεις διαφορετικές, αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχουν διαφωνίες. Όλοι προσπάθησαν να προσφέρουν το δικό τους λιθαράκι σε αυτό το οικοδόμημα που πρέπει να ε, οικοδομήσουμε και σε αυτές τις κοινέ αξίες που μας ενούν παρά τις πολιτικές μας διαφορές. Ποια λοιπόν είναι τα χαρακτηριστικά αυτών των τροπολογιών. σε ποια σημεία καλό θα ήταν να καταλήξουμε σήμερα σε συμβιβασμού, Σε συμβιβασμούς που κατά την άποψή μου είναι απαραίτητοι αν θέλουμε να μετριάσουμε κάποιε διαφορέ, αλλά κυρίω για να συνοψίσουμε, να ε, έχουμε μια πιο συνθετική παρουσία των τροπολογιών. Δεν μπορούμε να συμπεριλάβουμε 237 τροπολογίε. δεν πρόκειται να ε, λέγεται έκθεση αυτό το οποίο θα προκύψει. Όλη την εβδομάδα λοιπόν με τους σκιώδεις τρεις φορές ε, συνεδριάσαμε την Πέμπτη, θα συνεδριάσουμε για τέταρτη φορά, με στόχο να καταλήξουμε σε συμβιβαστικέ τροπολογίε που θα είναι πιο συνθετικέ, πιο συνεκτικέ και έτσι θα αποφύγουμε ε, κάποιε άλλε τροπολογίε. Ποια είναι τα πρώτα σημεία στα οποία θα ήθελα να επανέλθω. Πρώτα απ' όλα, ο ίδιος ο ορισμός της δημοκρατίας, αυτής της έννοιας που πραγματικά αξίζει να είμαστε στρατευμένοι στο στόχο της. Το ουσιώδες έχει γίνει νομίζω από την ομάδα Άλντε και από, από τον κύριο Λάμσντορφ. Μνημειώδες τα χαρακτήρισα το έργο το οποίο έχει επιτελέσει ο κύριος Λάμσντορφ ο οποίος έχει φανταστεί μια διαφορετική δομή για την έκθεση αυτή. Είχαμε μια διμερή επαφή στο Στρασβούργο. Η πρόταση του Λάνσντορφ ίσω να ήταν πιο ευφυή από αυτή που είχα εγώ σκεφτεί καταρχήν, που περιλάμβανε τρεις πτυχές. Αλλά αν είχαμε μπορέσει στο Στρασβούργο να συμφωνήσουμε οι δυο μας, ε, από τη στιγμή που άρχισαν να φτάνουν τροπολογίες από τις άλλες πολιτικές ομάδες με την αρχική δομή της έκθεσης καταλαβαίνετε ότι ήταν αδύνατον να δεχθώ μια άλλη δομή γιατί θα έπρεπε να ξαναφτιάξω από την αρχή την έκθεση. Προτείνω λοιπόν και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και με το συνεργάτη του κυρίου Λάμσντορφ και την ομάδα μου ε, το εξετάζουμε είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε λοιπόν είναι να συγκρατήσουμε όσα ήθελε να πει η Δημοκρατία ο συνάδελφος αλλά να τα εντάξουμε στην υφιστάμενη δομή της έκθεσης. Και νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Λυπούμε που δεν μπορούμε να είμαστε θα ίσω θα ήταν καλύτερο το αποτέλεσμα, αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω με μία άρδιν ε, αλλαγή τη δομή τη έκθεση, γιατί θα έπρεπε να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα δομή όλε οι τροπολογίες, κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Δεύτερο θέμα, στο οποίο πάνω δουλεύουμε σκληρά αυτές τις μέρες για να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες. Πρόκειται για τα διάφορα μέσα, ιδίω για το μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ορισμένοι διατύπωσαν την πρόταση να υπάρχει ένα λεγόμενο endowment for democracy, ένα αντίστοιχο ε, ταμείο, ε, πόρο σαν αυτόν που υπάρχει στις Ηνωμένε Πολιτείες. Θα σας δώσω κάποια στοιχεία. Όπως ξέρετε, στις τροπολογίες ε, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, μεγάλη ποικιλία απόψεων. Κάποιοι προτείνουν αυτό το Endowment for Democracy, κάποιοι άλλοι στις τροπολογίες τους λένε ναι, συμφωνούμε με αυτό, αλλά εάν δεν καταλήξουμε ε, σε τροποποίηση των εφιστάμενων μέσων. Και υπάρχει και η αρχική πρόταση που λέει να μην δημιουργήσουμε νέα εργαλεία, νέα μέσα, ας βελτιώσουμε τα ήδη υφιστάμενα, τα οποία αξίζουν και βελτίωση και καλύτερη χρηματοδότηση και μεγαλύτερη ευελιξία πολλές φορές τι τώρα θα καταλήξουμε να υιοθετήσουμε ως ε, ε, γραμμή στην ομάδα μας, αυτό είναι υπό μελέτη. Ίσως την πέμπτη να είναι έτοιμο. Υπάρχουν τα μέσα. Η στήριξη της δημοκρατίας μπορεί να γίνει μέσω του Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα, του μέσου αυτού, αλλά μέσω και των εμπορικών συμφωνιών, ε, συμφωνίες σταθεροποίησης, όλα αυτά τα μέσα. Υπάρχουν όμως ανεπάρκειες υπάρχει υποχρηματοδότηση, δεν υπάρχει μεγάλη συνοχή και συνεκτικότητα, δεν τα χρησιμοποιούμε ούτε τα υλοποιούμε συχνά αυτά τα μέσα, άρα εκεί πρέπει να γίνει επί της ουσίας δουλειά. Εάν λοιπόν δεν καταλήξουμε αυτά τα μέσα, αυτά τα εργαλεία, να τα καταστήσουμε πιο ευέλικτα και πιο προβλεπτικά θα έλεγα, και βλέπουμε στις αραβικές χώρες σήμερα τις διαδικασίες αυτές μετάβασης, δημοκρατικής μετάβασης, πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Αν δεν καταλήξουμε με αυτά τα εργαλεία σε βελτίωση, θα μπορούσαμε να προβλέψουμε αυτό το Endowment for Democracy, αλλά να εμπίπτει στην τακτική δημοσιονομική διαδικασία και να υπάρχει full parliamentary control, πλήρης κοινοβουλευτικό έλεγχος. Αν υπάρχει αυτό το Endowment for Democracy, θα πρέπει να ενταχθεί, θα πρέπει να εγγραφεί στον προπολογισμό, τον τακτικό και να υπάρχει, όπως είπα, πλήρης κοινοβουλευτικός έλεγχος. Θα πρέπει να δούμε σε τι συμβιβασμό μπορούμε να καταλήξουμε. Δεν είμαστε κατά αυτού του νέου μέσου που έχει πολλούς υπέρμαχους, κυριάστον, ε, θα αποφανθεί σύντομα από αυτό όπως γνωρίζουμε, αλλά εμείς λέμε ότι καλό είναι να ενισχυθούν τα ήδη φυστάμενα μέσα πρώτα απ' όλα. και θα με εξέπλησε το γεγονός να υιοθετεί στο Κοινοβούλιο νέα μέσα χωρίς να έχει καν ε, το δικαίωμα λόγου και κοινοβουλευτικού ελέγχου. Δεν νομίζω ότι είναι η λύση που θα μπορούσε να υποστηρίξει η Επιτροπή μας. Θα σας υποβάλουμε λοιπόν γρήγορα μέχρι την πέμπτη ίσως αυτή την συμβαστική πρόταση. Τρίτο θέμα τώρα εκδημοκρατισμός μέσω εμπορικών συμφωνιών. Εδώ δεν έχουμε τόσο μεγάλες αποκλήσεις μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων για το σύνολο των τροπολογιών που έχουν υποβληθεί επί του σημείου αυτού και εκεί προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μια συνοπτική πρόταση που θα περιλαμβάνει τις διάφορες αποχρώσεις. Δεν φαντάζομαι να έχουμε τεράστιες δυσκολίες. Τέταρτο θέμα. Τέταρτη θέση τροπολογιών. αποστολές εκλογικής παρατήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράγραφοι 14 και 15. Και εδώ υπάρχει μια ολόκληρη δέσμη τροπολογιών. Ήδη έχουμε καταλήξει σε συμβιβαστικές προτάσεις μαζί με τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Βέβαια, αυτό στο οποίο αποσκοπούμε είναι να συνεχίσουμε να έχουμε και να στηρίζουμε αυτές τις αποστολές, να έχουμε δηλαδή ένα πληρέστερο εκλογικό κύκλο το πριν της ε, αποστολής παρατήρησης των εκλογών, το κατά και το μετά. Τρία στάδια, τρεις φάσεις. Και βέβαια να υπάρχει και στήριξη εκ μέρους του Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, όλης τέλο πάντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την ολοκλήρωση των αποστολών, για τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η αποστολή και να στηρίζονται τα συμπεράσματα στο οποίο καταλήγουν οι αποστολέ παρατήρηση εκλογών. Γιατί πολλέ φορέ τα συμπεράσματα, οι συστάσει ε, λίγο πολύ ελαφριά αντιμετωπίζονται από τους διάφορους πολιτικούς φορείς. Εγώ θα παραδεχθώ το δικό μου σφάλμα. Service d'action extérieure sur υλοποίηση ε, των συμπερασμάτων των αποστόλων εκλογικής παρατήρησης. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε το Συμβούλιο να ευθυγραμμιστούμε πάνω σε συστάσεις αυτών των αποστολών παρατήρησης εκλογών, που τις περισσότερες φορές εκπονούνται από κάποιους ε, τεχνοκράτες, δεν έχουν ψηφιστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρόκειται για συστάσεις που πιστεύω ότι θα πρέπει να τις περάσουμε από κόσκινο, να τις εξετάσουμε εξονυχιστικά. Δεν μπορούμε να ζητούμε η ΕΕΔ, η κυρία Άστον, δεν ξέρω κι εγώ ποιο, να το στηρίξει αυτό χωρίς να έχει επικυρωθεί από ένα όργανο που έχει πολιτική νομιμότητα. Που δεν είναι κατά ανάγκη αυτή, αυτό το όργανο, αυτός ο φορέας η αποστολή εκλογικής παρατήρησης. Μιλάω για την ευθυγράμμιση με τα συμπεράσματα. Να πούμε, αν υπήρξε ε, νοθεία παραδείγματο χάρη, ε, φυσικά και δεν λέμε ότι θέλουμε να ελοποιήσουμε με τα αποτελέσματα, αλλά όχι να το εντάξουμε στα συμπεράσματα. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των συμπερασμάτων της αποστολής, ότι δηλαδή ήταν δημοκρατική ή δεν ήταν δημοκρατική η διεξαγωγή των εκλογών και τι πρέπει να κάνουμε με τις συστάσεις, αυτή την ε, μακροσκελή έκθεση που υποβάλλεται μετά την αποστολή. Εκεί ίσως υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορούμε να δεχθούμε και άλλα που δεν πρέπει να δεχθούμε. Κάποιοι συνάδελφοι σωστά λένε να διαγραφούν κάποια στοιχεία από αυτή την πρόταση. Πέμπτο θέμα. Πάντα στο πλαίσιο των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί τρίτο τμήμα του κειμένου που έχει να κάνει με τη στήριξη της κοινωνικής δυναμικής. Εκεί να σας πω την αλήθεια μου, περίμενα να αντιμετωπίσω του κόσμου τις δυσκολίες, αλλά όχι σε αυτό το σημείο, που μιλάει για τη στήριξη της κοινωνικής δυναμικής στις χώρες αυτές. Δεν ξέρω, μήπως ε, κάποιο πρόβλημα μεταφραστικό υπάρχει τι θα πει κοινωνική δυναμική, τι θα πει κοινωνικό κίνημα. Δεν είναι το ίδιο, τουλάχιστον στη γλώσσα μου είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Μιλάμε για κάποιες οργανώσεις νεολαίας, ή ε, αγροτών ή γυναικών που προσπαθούν να εμπνεύσουν την κοινωνία σε κάποιο βαθμό, για κάποια υπόθεση. Λέω ε, κάποια δίκτυα που μπορεί να ανταλλάσσουν συνταγές μαγειρικής ή είδη πλεξίματος ή μπορεί να είναι άλλες, άλλα δίκτυα ε, τα οποία ζητούν άλλα πράγματα. Παραδείγματο χάρη ε, Σουδάν τώρα, η γεφύρωση νότου-βόρειου, ε, νότου-βορρά. Υπάρχουν τέτοιου είδου πρωτοβουλίε. Ότι να πούν οι γυναίκε ότι κοιτάξτε, δεν μπορεί να υπάρξει η νευτική διαδικασία αυτή καθεαυτή, αλλά μπορούμε να αναλάβουμε κάποιε πρωτοβουλίε γεφύρωση κτλ. Για αυτά τα αυθόρμητα κινήματα μιλάμε. Για την οικοδόμηση μια εναλλακτική ε, σε διαφθαρμένα καθεστώτα. Που δεν είναι το ίδιο με το κοινωνικό κίνημα, που είναι κάτι άλλο. Είναι τέλος διαφορετικό το ένα από το άλλο. Κάποιοι συνάδελφοί μου, ιδίως από το ΕΛΚ και από την ΑΛΤΕ, ήθελαν να αντικατασταθεί στο κείμενο η πτυχή αυτή, η κοινωνική δυναμική, με τον όρο κοινωνία των πολιτών. Δεν είναι το ίδιο. Η κοινωνία των πολιτών, ναι, εντάξει, φυσικά. Είναι πάρα πολύ σημαντική η κοινωνία των πολιτών. Αν ο πληθυσμό με τα διάφορα στρώματα, ε, τις, τα διάφορα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά, ναι, φυσικά να διατηρηθεί όμως η κοινωνική δυναμική. Να αλλάξω κάποια πράγματα είμαι έτοιμη. Αν δεν αντιστοιχούν ακριβώς ε, στη μετάφραση ίσως που θα πρέπει να γίνει προς τα αγγλικά. Εντάξει, δεν θα πεθάνω κιόλα, έτσι. Έχω πέρασει κι άλλες τις καταστάσεις, αλλά ε, αυτό το πνεύμα, ε, το πνεύμα που διαπνέει αυτή, το τρίτο κομμάτι, το τρίτο τμήμα της έκθεσης θέλω να διατηρηθεί. Και δεν καταλαβαίνω γιατί το ΕΛΚ, η Άλντε ε, διαφωνούν. Ξέρω όλο αυτό το κίνημα των χριστιανικών συνεταιρισμών, των χριστιανικών συνδικάτων. Ξέρω πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι θέμα πολιτικό, αν είμαστε σοσιαλιστέ, χριστιανοί, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Μιλάω για κάποια ομάδα που ξαφνικά παίρνει μια πρωτοβουλία. Τι ήταν η αλληλεγγύη ήταν κάτι που ξεκίνησε και μετά πήρε έτσι ένα πολιτικό νόημα. κάτω από πολύ απολυταρχικά διεφθαρμένα καθεστώτα, όταν δεν υπάρχουν πολιτικέ εναλλακτικέ κάποια δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί το απολυτορχικό καθεστώ δεν αφήνει να γεννηθούν τέτοια ε, σε έχουμε ένα άλλο είδους, ε, μια άλλη αφύπνιση κάποιων ομάδων. Αυτό εννοώ όταν λέω κοινωνική δυναμική. Δεν ξέρω, πρέπει να βρούμε μια διατύπωση που να επιτρέψει να παραμείνει δι' αυτή στο κείμενο. Αυτοί είναι οι πέντε τομείς για τους οποίους σήμερα χάρη πραγματικά στην αξία οθαύμαστη συνεργασία των σχεδόν από όλες πολιτικές ομάδες, γιατί βέβαια δεν είναι μόνο, μάλλον να πω δε ότι δεν είναι μόνο οι σκιώδεις εισηγητές, έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και άλλοι συνάδελφοι. Δεν θέλω καν να τους κολακεύσω, ε, έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά και θα προσπαθήσω τον πλούτο των τροπολογιών τους να, την, να τον διατηρήσω. Αλλά χωρίς να τροποποιήσω εκ βάθρων την έκθεση για να κρατήσει την αρχική της, ε, το αρχικό της νόημα. Βεβαίως έχω μπροστά μου όλες τις τροπολογίες. Δεν θέλησα όμως να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Σας ε, παρουσίασα τη γενική οικονομία του σχεδίου έκθεσης που είναι πάρα πολύ σημαντικό Όλοι το περιμένουν, όλοι ε, το θεωρούν πολύ σημαντικό γιατί μιλάμε για ένα ζήτημα κεφαλαιόδους σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Grazie. Σας ευχαριστώ. Έχουμε τέσσερις παρεμβάσεις, πέντε. Ξεκινάμε με την συνάδελφο Χαουτάλα, πρόεδρος της Υποεπιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω ότι η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ σε έκθεση σημείο. Καταρχάς, το Συμβούλιο έχει δημοσιεύσει το Δεκέμβριο του 2009 τα σχετικά συμπεράσματα και επίσης θεωρώ ότι και οι εξελίξεις στον αραβικό κόσμο αποτελούν ένα λόγο για τον οποίο επιπλέον θα πρέπει να σκεφτούμε με προσοχή πώς θέλουμε να προωθήσουμε τη δημοκρατία. Όπως ανέφερε και η συγγήτρια, η Πολωνική Προεδρία και ο Πολωνός Υπουργός Εξωτερικών προωθεί ενεργά τα νέα οικονομικά εργαλεία για την προώθηση της δημοκρατίας σε τρίτες χώρες και συμφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι σωστές δομές μεταξύ άλλων και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Θα ήθελα τουλάχιστον τα μέλη που εργάζονται για την έκθεση αυτή, να συναντηθούν εκ των με την Πολωνική Προεδρία, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το σχέδιο και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει στην όλη διαδικασία. Ίσως θα υπάρξει κάποια δυνατότητα να εξετάσουμε ποιες είναι οι προκλήσεις και τα ελλείμματα σε ό,τι αφορά την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον εκδημοκρατισμό αυτή η νέα ευρωπαϊκή κληρονομιά για την δημοκρατία ίσως θα μπορούσε να αντικαταστήσει εν μέρη αυτό το εργαλείο. Εν πάση περιπτώσει να τα σκεφτούμε και τα δύο από κοινού. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι η συγγήτρια μας έχει παρουσιάσει τις, ε, σχέσεις, τις σκέψεις της για τις επιτροπές ε, παρακολούθησης των εκλογών, γιατί επί του παρόντος πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν εκτελούν πάντα το έργο τους και είμαστε υπεύθυνοι ως Κοινοβούλιο για τις αποστολές αυτές. Έχουμε και μία ομάδα εργασία με τον κύριο Αλμπερτίνη και την κυρία Ζολή ως Προέδρους. Θα έπρεπε να καθορίζουμε περισσότερο τη διαμόρφωση του έργου αυτών των ε, αντιπροσωπιών παρατήρησης των εκλογών. Θα πρέπει να υπάρχει μακροπρόθεσμος σχεδιασμό θα πρέπει να μην χρησιμοποιούνται ως πολιτικό εργαλείο όπως συμβαίνει πολύ συχνά σήμερα. Κάποιοι γελούν. Ελπίζω να μην γελούν μαζί μου. Η έκθεση λοιπόν αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει μια ευκαιρία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να επαναορίσει τις ε, τα κριτήρια των αποστολών αυτών. Θεωρώ ότι οι 237 τροπολογίες ουσιαστικά εμπλουτίζουν την έκθεση της συγκήτριας και είμαι βέβαιη ότι τελικά θα είναι πάρα πολύ συνεκτική η έκθεση όταν θα συζητήσει η συγγήτρια και με τους κοιόδης το τι σκοπεύει να κάνει. Χαίρομαι που οι συνάδελφοι έχουν καταθέσει πολλές τροπολογίες που συνδέουν το θέμα της δημοκρατίας με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτούμε χωρίς να υπάρξουν ε, αλληλεπικαλύψεις με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα μας δώσει η ΕΕΣ τον Ιούλιο. Και θα ήθελα να υπάρξουν κάποιοι, μου αρέσουν μάλλον κάποιοι από τους ορισμούς του κυρίου Κουκάν, αν δεν κάνω λάθος, για το τι είναι η δημοκρατία η 19 για παράδειγμα, η τροπολογία. Αυτό να το διαβάσουμε καλά, γιατί η δημοκρατία δεν περιλαμβάνει μόνο τις εκλογές. Άρα, να πω ότι πραγματικά θα ήθελα να υπάρξει αντίκτυπος ε, της έκθεσης αυτής στην τελική της μορφή. Bene, eh, la parola al collega Kukan. Purtroppo, purtroppo. Το λόγο είχε ο κύριος ε, Κούκαν. Προσθέθηκαν δε και άλλοι ομιλητές, γι' αυτό παρακαλώ να είστε σύντομοι. Δύο λεπτά έκαστος. Κύριος Κούκαν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλέ τροπολογίε κατέθηκαν για την έκθεση αυτή και αυτό καταδεικνύει το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για τον εκδημοκρατισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των εξωτερικών σχέσεων. Να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα το έργο της συγγύτριας και να ευχαριστήσω και τους ε, συναδέλφους για τις προσπάθειές τους και για τις ε, θετικές παρατηρήσεις τους. Όπως είπε η κυρία Καλτάλα, συζητούμε τις ε, πολιτικές αυτές σε μια χρονική συγκυρία όπου βλέπουμε ότι υπάρχουν τάσεις για πρόοδο προς την δημοκρατία σε πολλά μέρη του κόσμου. Ο εκδημοκρατισμός και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να τοποθετηθούν στο επίκεντρο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την εξωτερική διάσταση. Κάποιες τροπολογίες οι οποίες ε, θέτουν σωστές προτεραιότητες για την έκθεση αυτή. Επιτρέψτε μου να αναφέρω η τροπολογία που καλεί για το mainstreaming την, στο συντονισμό των πολιτικών εκδημοκρατισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενισχύει τη διαδικασία ε, διεξαγωγής διαλόγων, διαλόγου. Στο σημείο αυτό θα ήθελα επίσης να τονίσω το εξής. Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση στην Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της προσοχής μας, δεν θα πρέπει η προσέγγιση μας να βασιστεί μόνο στις δύο αυτές περιφέρειες. Χρειάζεται υποστήριξη από πλευρά μας, όχι μόνο σε υποθέσεις ανερχόμενων, ανδιόμενων δημοκρατιών. Χρειάζεται μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση για όλες τις χώρες που περνούν μέσα από μια διαδικασία εκδημοκρατισμού. Να μην ξεχνάμε ότι και τα νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν καλές εμπειρίες σε ό,τι αφορά τη διαδικασία εκδημοκρατισμού. Καλή ιδέα θα ήταν, θεωρώ, επίσης να υποστηρίξουμε τις τροπολογίες μας, τις τροπολογίες που έχει καταθέσει ο συνάδελφος Λάμσδορφ, 1.31.45. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε να βρούμε ένα γενικό ορισμό του εκδημοκρατισμού, αλλά θα ήταν ωφέλιμο να προσπαθήσουμε να ορίσουμε κάποια βασικά στοιχεία στην έκθεση σε ό,τι αφορά τα εργαλεία εκδημοκρατισμού, πολλές ε, τροπολογίες κινούνται προς την ίδια σωστή κατεύθυνση. Υποστηρίζω τις τροπολογίες που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Κληρονομιάς. Και τέλος, Πρόεδρε, Νομίζω ότι το τελευταίο τμήμα θα πρέπει να επικεντρωθεί στα κινήματα της κοινωνίας των πολιτών και θα πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν την υποστήριξή μας προς τις οργανώσεις αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο άλλος και ο δισηγητής, ο κύριος Λάμπστορφ. Ευχαριστώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω την Περονίκ που ήταν τόσο επικοδομητική καθ' όλη τη διαδικασία αυτή. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι είμαι πολύ ευτυχής που θέλει να συμπεριλάβει μία απόπειρα ορισμού ίσως της δημοκρατίας, αλλά ίσως όχι, ίσως μία κοινή ε, συμφωνίας για το τι περιέχει μια πραγματική βιώσιμη δημοκρατία. Θα πρέπει να υπάρξει κάτι τέτοιο και θα πρέπει να συμφωνήσουν και τα άλλα θεσμικά όργανα. Άρα θεωρώ ότι με τον τρόπο αυτό προωθούμε την ε, ευρωπαϊκή συζήτηση. Αύριο θα δούμε και την έκθεση EMP του Επιτρόπου Φιούλε σε ό,τι αφορά και τον εκδημοκρατισμό. Μου προκάλεσε έκπληξη επειδή υποτίθεται ότι υπάρχει και ένα μέσο για την κοινωνία των <laughs> πολιτών και θέλουμε να διατηρηθεί αυτό το μέσο. Να ρωτήσω την Πολωνική Προεδρία να ζητήσω και από την Επιτροπή, να ζητήσω και από την ε, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να μας δώσουν μια συνεκτική και εναρμονισμένη προσέγγιση για όλα αυτά τα εργαλεία, γιατί ιδάλλως θα καταλήξουμε ε, με διαφορετικά μέσα στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, για παράδειγμα, αντικρουόμενα. Όλα τα, μέσα αυτά θα έχουν καλούς σκοπούς, αλλά θα είναι αντιφατικά τελικά. Άρα, εντάξει, είμαι υπέρ τη Ευρωπαϊκή Κληρονομιά για τη Δημοκρατία, το έχω συζητήσει σε πολλέ ευκαιρίε αυτό το θέμα, είναι καλή ιδέα καλό μοντέλο, αλλά θέλω να υπάρχει συστηματικός ορισμός για το τι θέλουμε να πετύχει η κοινωνία των πολιτών, πώς σχετίζονται όλα αυτά τα μέσα και πώς θα δαπανιστούν τα κονδύλια αυτά. Θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει ήδη σχέδιο συνθήκης που έχει διανεμηθεί, θα πρέπει να το εξετάσουμε. Και σε ό,τι αφορά τις αποστολές παρατηρήσεις εκλογών, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για την κοινωνική δυναμική. Θεωρώ ότι ίσως αυτό να αποτελεί γλωσσικό θέμα. Θεωρώ ότι η κοινωνία των πολιτών έχει να κάνει με αυτά που λέτε, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε συμβιβασμό προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Bene, allora, agli altri... Μάλιστα. Υπόλοιποι συνάδελφοι. Χρειασμένοι ένα λεπτό για κάθε παρέμβαση, λυπούμε, αλλά υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα όρια. Συνάδελφος Τζάλα. Ευχαριστώ. Να πω ότι συμφωνώ με την προσέγγιση της εισηγήτριας και όλοι συμφωνούμε ότι στο σημείο αυτό είναι πολύ σημαντική η χρονική συγκυρία. Η κατάσταση έχει αλλάξει. Στο παρελθόν η διαδικασία εκδημοκρατισμού ήταν μια απόπειρα ε, επιρροή στις ε, ελίτ και στις κυβερνήσεις. Πλέον υπάρχει, υπάρχουν πολύ ε, μεγάλα κοινωνικά κινήματα και θα πρέπει να προσαρμοστεί και η προσέγγιση μας στην αυτή η πραγματικότητα. Και μετά από τη ζημιά που προκλήθηκε ιδιαίτερα από την, προ, την, τις μεθόδους του της πρώην κυβέρνησης Μπούς σε ό,τι αφορά την διαδικασία εκδημοκρατισμού. Θα πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή λοιπόν και η έκθεση αυτή περιλαμβάνει κάποιες προτάσεις και γι' αυτό συμφωνώ ιδιαίτερα με την πρόταση. Thank you for the ε, Το λόγο έχει η Συνάλφος Γκόμες. Ένα λεπτά. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ συγχαίρω τη Βερονίκη για την ε, εργασία της και την ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό για τις σχέσεις που θέλουμε να αναπτύξουμε με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου. Εγώ μόλις έρχομαι από τη Λιβύη και το μήνυμα είναι πολύ σαφές. Καταλαβαίνω τι, τι θέλει να πει η Βερονίκ για την κοινωνική δυναμική, γιατί αυτό ακριβώς βλέπουμε για παράδειγμα στη Λιβύη όσον αφορά τον έλεγχο της αρχής του Τένσε. Η ΜΚΟ ε, εκρήγνεται. 60 ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το περιβάλλον και ούτω καθεξής, αλλά χρειάζονται πάρα πολύ capacity building και αυτό ακριβώς μας ζητούν. Σύμφωνα επίσης με τα κριτήρια για τα θέματα αποστολών παρατήρησης των εκλογών, πιστεύω ότι θα πρέπει να πούμε στην ύπατη εκπρόσωπο ότι δεν μπορεί να προτείνει αποστολές εκεί όπου δεν παρακολουθήσαν τις δικές μας συστάσεις. Σημαίνει δηλαδή ότι αυτές οι κυβερνήσεις δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για τη μετάβαση στη δημοκρατία. Θέλουν μεν τον, την πολιτική εξοπιστία μπορούμε να τους δώσουμε, στέλνοντας αποστολές παρατήρησης τώρα. Για τα υπόλοιπα θέματα συμφωνώ ότι αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, το χρειαζόμαστε είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να σχηματιστούν ε, πολιτικά κόμματα, γιατί δεν υπάρχουν εκλογές χωρίς πολιτικά κόμματα και άρα όντως θα πρέπει να βοηθήσουμε, αλλά ε, πρέπει να είναι υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως εξάλλου συμβαίνει με το Αμερικό endowment ε, για τη δημοκρατία υπό τον έλεγχο του Κογκρέσου. Σάιρους και παρακαλώ. First, να ξεδιευκρινίσω κάποια πράγματα και να απαντήσω και κάποιες ερωτήσεις της συναδέλφου Ντεκέιζερ. Καταρχάς, ε, δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει άλλα μέσα αυτή η Ευρωπαϊκή Κληρονομιά για τη Δημοκρατία, γιατί δεν είναι το εκτελεστικό όργανο που θα διδάξει τη δημοκρατία. Θα πρέπει να υπάρχει κοινοβουλευτική εποπτεία. Το δεύτερο θέμα θα πρέπει να είναι συμπληρωματικό προς αυτά που υπάρχουν. Και από πλευρά κονδυλίων θα πρέπει να αφαιρέσει κονδύλια από ήδη υφιστάμενα μέσα. Δεν θα πρέπει, θα πρέπει μάλλον να θέσει μια στρατηγική. Μιλάμε για 100 ε, εκατομμύρια ευρώ. Παρόμοιο ποσό με αυτό που δίνεται στο αμερικανικό αντίστοιχο μέσο. Θα πρέπει να επικεντρωθεί στα κόμματα, στα κοινοβούλια, προκειμένου να αντικατασταθούν αυτά που υπάρχουν σε ολιγαρχικές κοινωνίες. Θα πρέπει να είναι αποκεντρωμένα από πλευράς χρηματοδότησης, θα πρέπει δηλαδή η ιδιοκτησία να είναι στα χέρια των κομμάτων, των εργοδοτών, των συνδικάτων, των οργανώσεων, ακαδημαϊκών και το καθεξήν. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν αποκέντρωση της πολιτικής μας για να δοθεί χρηματοδότηση σε αυτές τις ομάδες, οι κοινωνικές, στις χώρες τις οποίες έχουμε στο στοχαστρό μας. Το 50% θα πρέπει να δαπανάτε για τα πολιτικά κόμματα και τα ιδρύματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα υπόλοιπα στους εμπλεκόμενους φορείς. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν και πρέπει να υπενθυμίσω ότι είμαι ο σκιώδης συζητητή εκ μέρους της ΓΚΟΕ και περιμένω μια ανοχή στο χρόνο, ίσως και στη σειρά των ομιλητών. Το θέμα που συζητάμε είναι πολύ σοβαρό. Η δουλειά που έχει κάνει η εισηγήτρια είναι σε πολύ θετική κατεύθυνση. Δεν πέφτει στον πειρασμό να συνεχιστεί η αντίληψη ότι η δημοκρατία εξάγεται. Η δημοκρατία δεν εξάγεται. Αυτό είναι το πικρό συμπέρασμα που βγάζουμε και από τις τελευταίες εξελίξεις και κινείται με δημοκρατική ευαισθησία στην έκθεσή της με την οποία συμφωνούμε. Επειδή ο χρόνος έχει περάσει, θέλω τρία σημεία γρήγορα στα οποία έχουμε κάποιες επιφυλάξεις ή και δεν τα βλέπουμε με τον τρόπο που βλέπονται είτε οι τροπολογίες είτε σε κάποια σημεία της έκθεσης. Η έκθεση κινείται, ξαναλέω, σε θετική κατεύθυνση. Το πρώτο, σε πολύ χοντρές γραμμές, πρέπει να έχουμε αίσθηση των ορίων της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι το ξεπέρασμα αυτών των ορίων μας δείχνει ότι πρόκειται περί παρεμβάσεων μέσα στις εξελίξεις κάποιων χωρών και μάλιστα με κριτήρια όχι πάντα την υπεράσπιση της δημοκρατίας και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η δεύτερη παρατήρηση είναι σε σχέση με τη χρηματοδότηση των πολιτικών δυνάμεων και των πολιτικών κομμάτων και αναφέρομαι σε σχετικές τροπολογίες παρότι μπορεί να θέσει κανείς θεωρητικά κάποια κριτήρια αντικειμενικά, πολλές φορές αυτή η διαδικασία χρησιμοποιείται για παρέμβαση και μεροληπτική υποστήριξη ορισμένων πολιτικών δυνάμεων. Με αυτή τη λογική θα έχουμε την ευκαιρία να το ξανακουβεντιάσουμε. Είμαστε αντίθετοι με ιδρύματα τύπου Δημόκραση. Ναι, το, το αυτό. Και το τρίτο, είναι ο ορισμός της δημοκρατίας. Θα έλεγα μια γενική σκέψη, αυτές οι πολιτικές έννοιες, όσο προσπαθείς να ψάξεις να βρεις τον τέλειο ορισμό, μάλλον στο τέλος καταλήγεις σε λάθος. Η δική μας η άποψη είναι, διότι δεν πιστεύουμε πως η Επιτροπή μας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ, να μείνουμε στον ορισμό της απόφασης του ΟΗΕ. Ευχαριστώ πολύ και θα έχουμε την ευκαιρία. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Τελείωσα και η συγγήτρια έχει δείξει τη διάθεση ότι μπορούμε να κάνουμε καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ehm. Ευχαριστώ. Είχατε το χρόνο που δώσαμε και στους κοιόδης εισηγητές και λίγο παραπάνω. Αλλά ε, νόμιζαμε ότι ήταν η συνάδελφος Βερζά, Βερζά ε, ως ε, σκιώδης για αυτή την έκθεση. Η κυρία Μουνής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Ντεκεζέρ για την εξαιρετική έκθεση που μας παρουσίασε πολύ επίκαιρη και κυρίως αντικατοπτρίζει τη δημοκρατική ευαισθησία της εισηγήτριας αλλά και των σκιωδών εισηγητών μέσω των τροπολογιών τους. Ένα από τα βασικά σημεία της έκθεσης που αφορά τις αποστολές παρατήρησης εκλογών, ένα θέμα πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο, που έχει δηλαδή με το μέσο αυτό μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο το Κοινοβούλιο, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να ενισχύσουμε και να διατηρήσουμε την νομιμότητα και την αξιοπιστία αυτών των αποστόλων παρατήρηση εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομιμότητα και αξιοπιστία που κερδίζονται με την καλή οργάνωση και καλή λειτουργία των αποστόλων παρατήρηση εκλογών, που σίγουρα επιδέχονται περαιτέρω βελτίωση, αλλά ήδη έχουν διανύσει μακρά διαδρομή, έχουν ένα κύρος και ένα γόητρο σε διεθνές επίπεδο και βέβαια μπορούμε να το πετύχουμε αυτό και με την παρουσίαση εκπροσώπων των πολιτών. Δηλαδή βουλευτές να πηγαίνουν στις αποστολές παρατήρησης εκλογών. Νομίζω ότι πρέπει να φροντίσουμε να διατηρηθεί το στοιχείο αυτό και αν προταθεί κάποιο είδος συμμετοχή ατόμων που δεν είναι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτό να γίνεται στο περιθώριο των αποστόλων παρατήρησης εκλογών και σε καμία περίπτωση ως μέλη της αποστολής παρατήρησης εκλογών του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Τελευταία παρέμβαση. Συνάδελφος Ζιμπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Dobrych słów, które mówią o kształcie. Ευχαριστώ. Και εγώ συμφωνώ με όλα τα καλά λόγια που ακούσαμε ήδη σήμερα για την έκθεση της κυρίας Δεκάιζερ. Από την πρώτη παρουσίαση στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η έκθεση αυτή έγινε πολύ καλά δεκτή. Εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι τα λεπτά ζητήματα τα οποία αναφέρονται στις τροπολογίες επίσης έχουν συνταχθεί σωστά και θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε συμβιβαστικές λύσεις. Εγώ είμαι ένας εκ των τριών συντακτών των τροπολογιών που φορούν το ειδικό ταμείο για τη δημοκρατία. Ε, πραγματικά πιστεύω πως αυτό το ταμείο θα πρέπει να υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Είναι απόλυτα φυσιολογικό το κοινοβούλιο να ασκεί έλεγχο και εποπτεία σε ένα τέτοιο κονδύλι, ε, πρικοδότηση. Και νομίζω ότι από τη μέχρι τούδη συζήτηση μπορούμε να καταλήξουμε στο ότι και εδώ θα είναι δυνατόν να φτάσουμε σε μια συμβιβαστική λύση. Εγώ είμαι πεπισμένο ότι η εμπειρία από τις πρόσφατες αλλαγές στη Βόρεια Αφρική είναι τέτοιου είδους που καταδεικνύει την ανάγκη ύπαρξης ενός τέτοιου ταμείου, γιατί ποιος θα μπορέσει να είναι έτοιμος να αναλάβει την κυβέρνηση εκεί, ενώ λείπουν τόσες υποδομές, λείπουν τόσα πολιτικά κόμματα, ιστός, θα είναι πολύ δύσκολο. Τέλος, το τελευταίο μου παρατήρηση αφορά τι καλές πρακτικές οι οποίε θα πρέπει να διαδοθούν, ιδιαίτερα αυτέ που προκύπτουν από την εργασία του διαμεσολαβητή, του Ombudsman. Ευχαριστώ. Τέλος, πέντε λεπτά, στην εισηγήτρια κυρία Ντεκεζέρα. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω την κυρία Χάουταλα και σημειώνω τα όσα μου είπε. Εγώ εκτίμησα ιδιαίτερο τι τροπολογίε τη και πιστεύω πω έχει δίκιο που υπογραμμίζει τη σχέση ανάμεσα στην δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κύριε Κούκαν, επίσης αναφέρατε, έχετε κάνει μια σειρά από τροπολογίες, δεν θα τι αναλύσω τώρα. Τι εκτιμώ πάρα πολύ επίση. Δεν ξέρω αν είχαμε την ευκαιρία να δούμε τον ε, βοηθό σας ή το, αν ήταν στο σύνολο των ε, βοηθών με τους οποίους ήρθαμε σε διαβούλευση. Ναι, είχε έρθει. Εντάξει τότε λοιπόν. Και εγώ ίδια θα είμαι στη συνεδρίαση της Πέμπτης, οπότε θα μπορέσουμε να το ξανασυζητήσουμε. Να Συμφωνώ με την ιδέα ότι η δημοκρατία, ο δημοκρατισμός είναι μια πολύ μακρόπνοη εργασία και πιστεύω πως και η ανακοίνωση που θα κάνει κάθε Άστον για την αναθεώρηση της πολιτικής γετνίασης ε, θα αναφέρεται σε αυτή την εργασία την μακρόπνοη και επιμένει σε αυτό. Εσείς μιλήσατε για την ιδέα του Ταμείου για τη Δημοκρατία και ο κύριος Γκζίμπ το ίδιο. Εγώ η ίδια πηγαίνω στη Βαρσοβία αύριο και θα έχω επαφές με την Πολωνική Προεδρία. Το λέω και προς τον κύριο Σάιρος Βόλσκι. Εγώ θα αναφέρω λεπτομερώς ε, τα όσα είπαμε, αλλά και θα λάβω υπόψη μου τη θέση της Προεδρίας. Είναι βασικά δύο πράγματα τα οποία μας ε, ε, δημιουργούν κάποια σύγχυση. Ε, ο κύριος Βόλης και ανέφερε την ανάγκη για κοινοβουλευτικό έλεγχο. για την ώρα δεν βλέπω την παραπληρωματικότητα. Φοβούμαι ότι θα υπάρξει επικάλυψη ή πάυση κάποιων ε, μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως το μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν πιστώ ότι θα είναι παραπληρωματικά και χρήσιμο ένα τέτοιο ταμείο, φυσικά και δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα για κάτι τέτοιο. Αλλά χρειάζονται περισσότερες ευκρινήσεις. Δεν είναι κάτι το πολύ εύκολο. Για τον κύριο Λάμστορφ απίδησα εν μέρη για το μέσο για τη δημοκρατία και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για το θέμα της κοινωνίας των πολιτών είμαι βέβαιο, βέβαιη ότι θα συμφωνήσουμε από αυτού. Δεν νομίζω πως είναι δυνατόν να αποτύχουμε. Για τον συνάδελφο Ζάλα επίσης ήδη έχω πει στον ε, βοηθό του πόσο εκτίμησα τις ε, τροπολογίες του που έχουν ένα διαφορετικό τόνο, διαφορετική χρειά. Στον κύριο Βόλκης, ε, Βόλκη απέντησα για τον κύριο Χουντή. Να σας πω ότι σίγουρα έχουμε διαφορές, όχι όμως για την τροπολογία σας 61 που θυμίζει το αναπαλωτρίο το δικαίωμα των λαών για την, στην αυτοδιάθεση και στην επιλογή της ε, δικής τους, ε, του δικού του είδους πολιτικής ανάπτυξης και διακυβέρνησης χωρίς εξωτερική παρέμβαση. Και μάλιστα θα το βάλω στην αρχή της έκθεσης και όχι εκεί που το τοποθετήσατε εσείς αν συμφωνείτε και για αυτό το σημείο φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε δεν είμαι απόλυτα σύμφωνη με τη, τη θέση της κυρίας Μονής, αλλά το έχουμε ήδη συζητήσει και πιστεύω πως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία των παλαιότερων συναδέλφων ευρωβουλευτών στις αποστολέ παρατήρησης εκλογών. Νομίζω πως έχουν, υπάρχει εμπειρία και η Μαρία Μονής μου είπε ότι δεν υπάρχει πλέον η δυναμιμότητα που έδινε παλιότερα μια τέτοια αποστολή παρατήρησης δεν δίνουμε το ίδιο κύριο, ίσως και ίσως με βεβαιότητα, αλλά ίσω να καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εμπειρία. Εγώ ήρθα σε επαφή με τον κύριο Πατ Κόξ, πρώην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά είναι σαφές ότι αν δεν θέλουμε απλώς να είναι μια φωτογραφία της κατάστασης, αλλά να υπάρχουν πραγματικά επιτόπου ευρωβουλευτές να ελέγχουν τι γίνεται στην κάθε χώρα και να πλαισιώνουν την κατάσταση, οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε και να μείνουμε επιτόπου για πολύ μεγάλο διάστημα. Θα μπορούσαν να το αναλάβουν οι πρώην βουλευτές, γιατί όχι. Μπορούμε να βρούμε λύσεις σε αυτό το επίπεδο. Κύριε Ξύμπ, ναι, ξέρω πως δεν λέω σωστά το όνομά σας. Σας ζητώ συγγνώμη. Κάνατε μια σειρά από τροπολογίες που μας ε, καλεί να μην ε, ξεχνάμε την Ανατολική Ευρώπη. Δεν την ξεχνάμε. Έχετε επιμείνει στις τροπολογίες σας. Είναι αλήθεια ότι η έκθεσή μου εστιάζεται στα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης. Αν και δεν αναφέρω ονόματα ούτε χώρες, αλλά έχετε δίκιο ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τις χώρες που είναι υπομετάβαση ή που βρίσκονται ακόμα υπό αυταρχικά καθεστώτα προς Ανατολάς και αυτές θα πρέπει να απελευθερωθούν οι χώρες. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Για μένα αυτό είναι τμήμα του συνόλου του προβλήματος και πιστεύω μάλιστα ότι η αναθεώρηση της πολιτικής συγκεκρινήσης δεν θα κάνει διάκριση μεταξύ Δύσης και Ανατολής και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις εμπειρίες μας για να βοηθήσουμε τους άλλους που ζουν σε άλλα πολιτικά πλαίσια. Ευχαριστώ. Νομίζω μίλησα λιγότερο για πέντε λεφτά. Εν πάση περιπτώσει, την Πέμπτη, το δεκάμιση με 1.30 θα έχουμε νέα συνάντηση με προτάσεις συμβιβαστικές για κάθε ένα από τα σημεία που αναφέραμε. Φυσικά, θα μπορούμε να τα ξανατροποποιήσουμε την Πέμπτη το απόγευμα. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Αντεκεζέρ. Επόμενο σημείο τώρα είναι το 10. Απολογισμό τη επίσκεψη αντιπροσωπεία για τη σχέση με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο τη στην και τη Δυτική Όχθη. Επίσκεψη που έγινε 26 με 28 Απριλίου του 2011 μέσα σε ένα πλαίσιο εξαιρετικά σημαντικό πολιτικό με την ανακοίνωση της ε, συμφιλίωσης ανάμεσα στις δύο βασικές ε, παλαιστινιακές ε, δυνάμεις και ενδυνάμωση του Παλαιστινικού Συντάγματος. Πριν να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Ντερόσα, θα ήθελα να καλωσορίσω και τον Γενικό Αντιπρόεδρο της, της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, της κυρίας Αλγασμίτου, που θα συμμετέχει στη συζήτηση ως ειδική επεσταλμένη της ΥΠΑ της εκπροσώπου. Έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας και γι' αυτό δίνω αμέσως στο λόγο στον συνάδελφο Ντερόσα. Παρακαλώ. Thank you very much, uh, Chair. Um, and thank you also. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση για να σας κάνω την παρουσίαση αυτή. Ήμουν πρόεδρος της αντιπροσωπείας αυτής από την αρχή της θητείας το 2009 και ήταν η πρώτη ευκαιρία που είχα να κάνω μια παρουσίαση στην Επιτροπή Εκτορικών Υποθέσεων, την οποία και εκτιμώ ιδιαίτερα. Καταρχάς, να ξεκινήσω λέγοντας και είμαι βέβαιος ότι η κυρία Έλγα Σμιτ θα το αναφέρει αυτό. Θα ήθελα να καλωσορίσω την δήλωση του Συμβουλίου, τη χθεσινή για το θέμα της Παλαιστινιακής Ισραηλικής, Ισραηλικής, Ισραηλινής ε, Ειρήνης. Ένα μια δήλωση για τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υπογραμμίσω ιδιαίτερα την παράγραφο 10 όπου αναφέρεται ότι θα υπάρξει συνεργασία με την ενδιάμεση κυβέρνηση, την υπηρεσιακή κυβέρνηση, την οποία προτείνει ε, θα προταθεί στην διαδικασία συμφιλίωσης. Τονίζεται επίσης η θέση στην παράγραφο 4 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία παρουσιάστηκε εκτενώς τον Δεκέμβρη του 2009 και επίσης να πω ότι χαίρομαι επειδή η Βαρόνι Άστον δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να ενεργοποιήσει το κουαρτέτο για να ανταποκριθεί στην τρέχουσα κατάσταση. Όπως αναφέρθηκε ήδη, η πρόταση αυτή περιλαμβάνει δύο Ιερουσαλήμ και ε, επίσης και το θέμα της Δυτικής Όχθης και έγιναν συζητήσεις με τα μέλη του PPLC, του PLC και με όλες τις ε, ομάδες και με κυβερνητικές ε, οργανώσεις της Παλαιστινιακής ε, Αρχής, του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου, επίσης με το γραφείο του ΟΗΕ για την Δυτική ε, όχθη και εδώ πέρα βλέπετε ε, μια έκδοση για τις ανθρωπιστικές ανησυχίες που επικρατούν για την Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως τις θεωρεί ο ΙΕΜ. Έγιναν συζητήσεις επίσης. Καταρχάς, μας υποδέχτηκαν οι επικεφαλής των αντιπροσωπιών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, που ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες μας σε ό,τι αφορά την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή. Έγιναν συζητήσεις με οικογένειες στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, ε, ιδιαίτερα με άτομα τα οποία είχαν εκδιωχθεί από τους απίκους. Ε, επισκεφτήκαμε τη Χευρώνα. όπου υπάρχει επαφή μεταξύ επίκων και των Παλαιστινίων πολιτών επισκεφτήκαμε ένα τζαμί, το οποίο επίσης ε, χρησιμοποιούν και οι, οι Εβραίοι της περιοχής ως ε, τόπο λατρείας. Κάναμε λοιπόν συζήτηση με τις οικογένειες αυτές, επισκεφτήκαμε το Ολκαρίμ, όπου συναντηθήκαμε με τις ε, τοπικές επιτροπές μη βίαιης αντίστασης αποτελούνται κυρίως από νέους που προσπαθούν να αποτρέψουν την βίαιη αντίδραση των νέων, να τους διοχετεύσουν σε ειρηνικές μορφές αντίστασης. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτόν, λαμβάνοντας υπόψη στο τι συμβαίνει και στην υπόλοιπη περιοχή. Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη. Προφανώς ε, οι Ισραηλινές ε, δυνάμεις ασφαλείας έχουν αντίκτυπο στην περιοχή και είδαμε ποιος ήταν ο αντίκτυπος αυτός. Και τα προβλήματα που δημιουργούνται σε ό,τι αφορά τις ταυτότητες στην Ιερουσαλήμ, για παράδειγμα, είδαμε οικογένειες, άνθρωπους, γυναίκες και άντρες που είχαν τους άντρες τους ή τις γυναίκες τους στην Βυτική Γάζα, αλλά επειδή δεν είχαν τα άτομα αυτά ταυτότητα Ανατολικής Ιερουσαλήμ, δεν μπορούσαν να τους επισκεφθούν εκεί. Και αν κάποιος ε, ε, επιλέξει να μείνει στην ε, Ραμάλα, δεν θα μπορέσει να κρατήσει την ταυτότητά του Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Υπάρχει και σχετική έκθεση του ΟΗΕ, την οποία σας καλώ να διαβάσετε. Τα συμπεράσματα από την επίσκεψή μας με ομοφωνία από πλευρά των μελών της αντιπροσωπείας από όλες τις ομάδες είναι τα εξή. Δεδομένη στις παράλυσης των ΗΠΑ στην ε, περιοχή αυτή επικρατεί η αντίληψη μεταξύ των Παλαιστινίων, των οποίων, τους οποίους συναντήσαμε, ότι ουσιαστικά το κουαρτέτο είναι νεκρό ως διαδικασία και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την εκκίνηση της όλης διαδικασίας. Αυτό καταδεικνύει την αξία της Ένωσης ως περιφερειακό φορέα, αν δούμε και την θετική στάση που κρατά ε, σε άλλες περιοχές, σε άλλες χώρες, στην ε, Λιβύη, στην Αίγυπτο και όλοι θεωρούν ότι πραγματικά ο χρόνος πιέζει πλέον. Ότι η διαρκής πίεση στους Παλαιστινίους, όχι μόνο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, αλλά και σε άλλα τμήματα της Δυτικής Όχθης, όπου όλοι, όλο και πιο πολλοί Παλαιστίνοι χωρίζονται από δρόμους, από επικισμούς Ισραηλινούς, κοιτώντας το χάρτη τώρα σε σχέση με το πώς ήταν και που βρίσκονται πλέον οι έπικοι θα δείτε μία σειρά αν θέλετε από που αντιπροσωπεύουν τις Παλαιστινιακές περιοχές που δεν ενώνονται μεταξύ τους και δεν λύνουν τα προβλήματα του τοπικού του κόσμου που μένει εκεί όπου μια διαδρομή 10 λεπτών μπορεί να πάρει 2 ώρες και τι θα πρέπει να περάσουμε και από σημεία ελέγχου κτλ. Υπάρχουν και τα πολιτικά προβλήματα στην Παλαιστινιακή περιοχή για το πώς θα δημιουργηθεί ένα βιώσιμο Παλαιστινιακό κράτος όταν είναι τόσο κατακαιρματισμένη η περιοχή. Αυτό το θέτω απλά και το καταθέτω απλά ως την άποψη των ε, ανθρώπων που ζουν εκεί. Αυτό που συμβαίνει είναι το εξής, όλοι το επιβεβαίωσαν. Είναι πραγματικά αδύνατον και αν δεν συμβεί κάτι σύντομα θα είναι πραγματικά αδύνατον να υπάρξει Παλαιστινιακό κράτος βάσει των ε, συνόρων του 67. Το ερώτημα είναι λοιπόν ποια θα ήταν η εναλλακτική λύση. Και φυσικά η εναλλακτική λύση θα ήταν ένα κράτος, ένα ενιαίο κράτος. Ποιος πιστεύει όμως ότι είναι βιώσιμη λύση το ένα ενιαίο κράτος. Πώς θα ζήσουν από κοινού σε βάθος χρόνου αυτοί οι δύο πληθυσμοί. Στην Ανατολική Ιερουσαλήμ η πίεση για την παιδεία, για παράδειγμα, είναι τεράστια λείπουν 1.300 τάξεις σχολείων. Υπάρχουν μεγάλες λήψεις σε ό,τι αφορά τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες είναι η υποπαλαιστινιακή διοίκηση σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών. Ανέφερα ήδη το πρόβλημα των επίκων. Όχι μόνο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ αλλά και στην Παλαιά Πόλη που δημιουργεί και τεράστια προβλήματα και στα σημεία ελέγχου. Τις πρώτες ημέρες της επίσκεψής μας ήμασταν αρκετά απεσιόδοξοι και την τρίτη ημέρα σε μία συνάντηση με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο μας διέκοψαν την συνάντηση για να μας πούν ότι είχε ε, Υπογραφή μια συμφωνία ε, επανασυμφιλίωσης στο Κάιρο. Είχαμε μόλις βγει από μια συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος μας είχε αναφέρει ότι γινόταν σχετική συνάντηση, χωρίς όμως ε, να μας πει ότι υπήρχε οποιαδήποτε ελπίδα για σύναψη συμφωνίας. Όλοι λοιπόν, σχεδόν όλοι από πλευρά του Νομοθετικού Συμβουλίου, χάρηκαν για την σύναψη της συμφωνίας αυτής. Και στη συνέχεια, όπου και να πήγαν, όπου και να πήγαμε, η ερώτηση που μας ε, θα ήταν διαρκώς ήταν πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναγνώριζε το αποτέλεσμα των εκλογών ή κατά πόσον θα αντιδρούσε όπως το 2006 και θα απέρριπτε το αποτέλεσμα μετά από τα όσα συνέβησαν στην Τινησία, στην Αιγύπτο, δεν μπορούσαμε, δεν θα μπορούσαμε να προβλέψουμε μια κατάσταση κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα αναγνώριζε το αποτέλεσμα νόμιμων ανώθευτων εκλογών. Αυτό απάντησα και ελπίζω να μην έκανα λάθος. Αυτή η αισιοδοξία που ξαφνικά επικράτησε ήταν πραγματικά απτή. Δεν άλλαξε όμως τους όρους εργασίας τις συνθήκες εργασίας και όπως ε, αναφέρει και το, η σχετική διακήρυξη, η σχετική δήλωση του Νομοθετικού Συμβουλίου, η διαδικασία είναι υποπαράλυση. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει για να προωθηθεί η κατάσταση. Είναι σημαντικό αυτό ως δήλωση και είναι και σημαντική και δήλωση του Προέδρου Ομπάμα της προηγούμενης εβδομάδας. Ξέρω ότι υπάρχουν αρκετές επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά τους ε, επικισμούς, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει τη θέση που έχει λάβει, ότι θα πρέπει να προωθήσουμε και να σημειώσουμε πρόοδο σε όλα τα σημεία. Ο Υπουργός Εξωτερικός, τον οποίο συναντήσαμε, ο Παλαιστίνιος ε, Πρόεδρος, ε, ο Υπουργός Εξωτερικών, κατέστησε σαφές ότι ελπίζουν να σημειωθεί πρόοδο το Σεπτέμβριο στον ΟΗΕ με, τα, με τη συμμετοχή στον ΟΗΕ και ανέφερε με σαφήνεια ρητά ότι η ημερομηνία αυτή δεν ήταν κάτι το οποίο δεν θα δεχτούν να αλλάξουν. Αν υπάρχουν σοβαρά ζητήματα σε ό,τι αφορά τα σύνορα θα μπορούσε να μετατεθεί αυτή η ημερομηνία. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και αυτές οι πληροφορίες σίγουρα φαντάζομαι θα έχουν μεταφερθεί στα σχετικά εμπλεκόμενα μέρη. Θεωρώ όμως ότι αποτελεί μια σημαντική ένδειξη ότι υπάρχει ένας βαθμός ευελιξίας στο σημείο αυτό σε ό,τι αφορά την πρόθεση της όλης διαδικασίας, γιατί κανένας από τους Παλαιστινίους που γνωρίσαμε δεν πιστεύει ότι θα υπάρξει ειρήνη χωρίς διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ και ότι δεν θα υπάρξει, κανείς δεν είναι σίγουρος ότι θα υπάρξει ασφάλεια. Αλλά μας ζήτησαν να έχουμε υπόψη ότι και οι Παλαιστίνοι χρειάζονται ασφάλεια. Δεν μπορούν να συνεχίσουν να ζουν με την απειλή βομβαρδισμού. Και ότι η ειρήνη θα πρέπει να βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην αμοιβαία ασφάλεια. Αυτό ασφαλώς θα πρέπει να το έχουμε υπόψη. Να πω επίσης ότι, και κλείνω πρόεδρε, ότι άκουσα από μια έκθεση του Γαλλικού Πρακτορείου ότι ο ηγέτης της ΦΑΤΑ είπε ότι δεν σκοπεύουν να προχωρήσουν με μονομερή διακήρυξη ανεξαρτησίας. Μπορεί να υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτού και τη συμμετοχή στον ΟΗΕ, αλλά θα ήθελα στο σημείο αυτό να κλείσω διευκρινίζοντας δύο στοιχεία. Καταρχάς, είναι σημαντικό στις ε, τρέχουσες συνθήκες το Κοινοβούλιο να έχει ένα μηχανισμό για να παρακολουθεί τα όσα συμβαίνουν. Προτείνω, εγώ το έχω συζητήσει αυτό βέβαια με τον κύριο Πέτερινγκ ή με κανέναν άλλον, αλλά θα μπορούσε να δώσει εντολή η Επιτροπή ΑΦΕΤ στην ε, Ομάδα Εργασίας για την Μέση Ανατολή προκειμένου να παρακολουθεί την κατάσταση και να ενημερώνει την ΑΦΕΤ. Και θα είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο, θεωρώ, να κάνει και το ίδιο συζητήσεις για την ερευνητική διαδικασία τώρα και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την μεσέντολη. Ξέρω ότι υπάρχουν και άλλα θέματα πιο μεγάλα, αλλά θεωρώ ότι το ζήτημα αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους βουλευτές. Να υπάρξει μια συζήτηση ή να υπάρξει ίσως και ένα ψήφισμα που θα αποτυπώνει την τοποθέτησή μας. Και σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις με το κουαρτέτο, με τον ΟΙΕ, και στα πλαίσια της Παλαιστινιακής Αρχής. Πριν να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, νομίζω πως θα ήταν σκόπιμο να ακούσουμε τα όσα έχει να μας πει η κυρία Έλγα Σμιτ όσον αφορά την ενημέρωση για την κατάσταση στην περιοχή. Και μετά οι συνάδελφοι που θέλουν να παρέμβουν θα Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε και μου δώσατε έτσι τη δυνατότητα να μιλήσω για αυτό το θέμα. Θα ήθελα να απαντήσω σε αρκετά από αυτά που αναφέρθηκαν και να πω ότι συμφωνώ με πολλά σχόλια. Ένα σημείο για το οποίο δεν συμφωνώ και το λέω αυτής εξ αρχής είναι ότι το κουαρτέτο είναι νεκρό. Όχι, δεν είναι νεκρό. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για να το αναστήσει, αν θέλετε, εντό αγωγικών. Θα σας ε, εξηγήσω λίγο πιο διεξοδικά τι εννοώ. Νομίζω ότι καταφέραμε να ξαναλειτουργήσει το κουαρτέτο. Συνεδριάσαμε το Φεβρουάριο. Οπότε το εκπρόσωπο στο Μόναχο προείδρευσε και φιλοξένησε αυτή τη συνάντηση και ο στόχος τότε ήταν να έχουμε μια δήλωση, να καταλήξουμε σε μια δήλωση του κουαρτέτου που θα βοηθούσαν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και οι δύο πλευρές. Αυτό έγινε το Φεβρουάριο όταν είχαμε γεγονότα ε, στην Αίγυπτο και σε άλλες χώρες και θεωρήσαμε ότι είναι κατάλληλη χρονική στιγμή. Πράγματι, απεσταλμένοι του κουαρτέτου εκλήθησαν να έχουν ε, συναντήσεις με διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές, και την Ισραηλινή και την Παλαιστινιακή, για να δουν τι ε, χρειάζεται ώστε να επανέλθουν ε, στις διαπραγματεύσεις και οι δύο πλευρές. Υπήρξαν αρκετοί γύροι διαπραγματεύσεων με τους εκπροσώπους, ε, τους, με τους δύο διαπραγματευτές. Ήταν πάρα πολύ καλές οι συναντήσεις που είχαμε και στην περιοχή αλλά και στις Βρυξέλλες. Για πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δύο φορές χρειάστηκε να αναβληθεί η συνάντηση του κουαρτέτο, αλλά αύριο συνεδριάζει στο κουαρτέτο, στο Παρίσι, για να σας πω. Και θα δούμε και τις τελευταίες εξελίξεις και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και σίγουρα θα έχουμε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε αυτή την ορμή και την όθεση που έδωσε η ομιλία που αναφερθήκατε κι εσείς του Πρόεδρου Ομπάμα. Ήμουν στη Γόσιγκτον, μάλιστα μαζί ε, με την πατεκπρόσωπη την προηγούμενη εβδομάδα, ακριβώς πριν ε, την ομιλία του Ομπάμα ήταν και βασιλιάς της Ιορδανίας εκεί, κατά σύμπτωση, ήταν μια πολύ στρατηγική στιγμή και στάλει ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα, γιατί αυτό ήταν αναγκαίο. Και φυσικά και ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη ομιλία Ομπάμα και ιδίω σε ό,τι αφορά ε, τα σύνορα του 67 που πρέπει να τηρηθούν, ασφαλή σύνορα και για τις δύο πλευρές. Ε, επίσης διασκεδάζονται ανησυχίε του Ισραήλ για την ασφάλεια και βέβαια συμφωνεί για την Ανατολικά Ιεροσόλυμ και τους πρόσφυγες. Αναφερθήκατε και εσείς αυτά. Είχαμε και μια πολύ σημαντική συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων ε, τα συμπεράσματά του επιβεβαιώνουν τη θέση μας, η οποία είναι ότι ζητούμε να ξαναρχίσουν επιγόντως οι διαπραγματεύσεις. Εσείς αναφερθήκατε στο Σεπτέμβριο. Είπατε επίσης ότι οι Ισραηλινοί είπαν ότι η προθεσμία του Σεπτεμβρίου ε, δεν είναι μια μετακίνητη ημερομηνία. Ακριβώς το ίδιο μας είπε ο επικεφάλης των διαπραγματεύσεων. Και όπως εκτιμούν τα πράγματα, αν Έχουμε διαπραγματευτική διαδικασία μέχρι το Σεπτέμβριο. Δεν χρειάζεται να γίνει και η Γενική Συνέλευση. Αυτή είναι η φιλοδοξία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των άλλων εταίρων του Κουαρτέτ να βοηθήσουν τι δύο πλευρέ να καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματεύσουν. Νομίζουμε ότι αυτό είναι απαραίτητο και γιατί υπάρχουν και πολλά ζητήματα τα οποία μπορούν να επιληθούν μόνο με τις διαπραγματεύσεις. Δεν αφορά αυτό το, μόνο την ασφάλεια, αλλά και άλλα ζητήματα πολύ σημαντικά, το νερό, τον ηλεκτρισμό και άλλα. Καταστήσαμε επίσης σαφές ότι αποθαρρύνουμε την λήψη μονομερών μέτρων ή επικισμή παραδείγματος χάρη από πλευράς Ισραήλ. Το έχουμε πει και επαναλάβει πολλές φορές στα συμπεράσματα του Συμβουλίου και στις άμεσες επαφές και συνομιλίες που έχουμε. Είναι παράνομοι οι επικισμοί και δημιουργούν εμπόδιο στην ειρήνη. Το είπε και είπατε εκπρόσωπος χθε στη δήλωσή της ε, μπροστά στα μέλη του τύπου. Ε, βέβαια αποθαρρύνουμε τις ε, μονομερείς ε, κινήσεις γιατί ενθαρρύνουμε ε, την ε, διαπραγμάτευση, τις διμερείς ε, προσπάθειες. Ανακοινώθηκε λοιπόν και η συμφωνία μεταξύ των διαφόρων φρατριών ε, της Παλαιστίνης και βέβαια εμείς πάντοτε ζητούσαμε να υπάρχει αυτή η Παλαιστινιακή Επανένωση υπό τον πρόεδρο Αμπάς ε, και γι' αυτό μας ε, ενθαρρύνει ιδιαίτερα η δήλωση του Καΐρου. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη δικρατική λύση. Βέβαια καταλαβαίνουμε ότι οι πλευρές συμφωνούν στην αρχή της Αποφυγή τη βία και δεσμεύονται να τηρήσουν τις προηγούμενες συμφωνίες και δεσμεύσει τους, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα του Ισραήλ να υπάρχει, το δικαίωμα ύπαρξης του κράτους Ισραήλ. Ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί είπατε για, για το ταξίδι μας Νομίζω ότι οι Παλαιστίνοι αναγνωρίζουν ότι εμείς είμαστε ο πιο σταθερός, αξιόπιστος ε, εταίρος. 500 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο παρέχουμε στην Παλαιστίνη από τον ε, προϋπολογισμό και μέσω του Ούνρα στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες και βέβαια μέσω διμερής οδρούς βοήθειας από τα κράτη-μέλη. Θέλω να πω όμως και κάτι ακόμη. Είμαστε στην πρώτη γραμμή και για, την, τη Γάζα. Ξέρουμε ότι η κατάσταση παραμένει ανησυχητική στη Γάζα. Είπατε εκπρόσωπος που πήγε εκεί, μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών, ήδη είναι η δεύτερη της επίσκεψη και έχουμε ζητήσει αλλαγή πολιτική στη Γάζα. Όχι μόνο για να περνάει ανθρωπιστική βοήθεια, ζητούμε άνοιγμα, αλλαγή πολιτικής. Κάτι τέτοιο θα επιτρέψει στη Γάζα να έχει τις ε, συναλλαγές, ε, τις κανονικές και βέβαια και εμπορικές ε, συναλλαγές και ανταλλαγές. Στηρίζουμε τους Παλαιστινίους, ιδίως ό,τι αφορά την αναβάθμιση των συνοριακών σημείων, των σημείων διέλευσης. Θα πρέπει οι Ισραήλ να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Έχουμε λοιπόν ένα κατάλογο μιλητών. Ο κύριος Ρόμπερτ Άτκινς είναι ο πρώτος ομιλητής. Πρόεδρε, έχω συμμετέχει σε δύο αποστολές ε, στην ε, Ιερουσαλήμ και την Παλαιστινιακή Αρχή υπό την ηγεσία του κυρίου Ντερόσα και τον συγχαίρω γιατί ήταν πραγματικά στο σωστό μέρος στη σωστή στιγμή. Μακάρι να ήταν και στις εκλογές στην ε, Βρετανία. Δεν έχουμε χρόνο να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες, αλλά να πω ότι τον υποστηρίζω και ξέρω ότι και άλλοι συνάδελφοι που έχουν συμμετάσχει σε ε, σχετικές αποστολές θα επιβεβαιώσουν τις ε, λεπτομέρειες. Ο δόκτωρ, η δόκτωρ Ασρά την προηγούμενη φορά που βρέθηκα εκεί μου δήλωσε ότι μας τελειώνει ο χρόνος. Βρισκόμαστε στο παραπέντε. Και αυτό είναι το σημείο το βασικό και το βασικό που θέλω να σας μεταφέρω ως μήνυμα. Είμαι σίγουρος ότι αυτό καταφέρει η Επιτροπή μας, το καταλάβει η Επιτροπή μας, αλλά δεν είμαι σίγουρος για το Κοινοβούλιο, είναι ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λάβει κάθε θετική δράση για να υποστηρίξει τη διαδικασία αυτή, δεν θα συμβεί τίποτα. Μας έχουν κατηγορήσει και το έχω ξανακούσει αυτό στο παρελθόν, μας κατηγορούν ότι πληρώνουμε, αλλά δεν είμαστε μεγάλοι ε, παράγοντες, payers και όχι players. Συμφωνώ και για το κουαρτέτο αυτό που είπατε. Οπουδήποτε και να πήγα, ε, το περιφερόν του κουαρτέτο. Θεωρούν ότι δεν έχει να παίξει οποιοδήποτε ρόλο και δεν θέλω να κάνω πολιτικό σχόλιο για τον κύριο Μπλερ εδώ πέρα. Αλλά εμείς και μπορούμε και πρέπει να δράσουμε. Και αυτό που με ανησυχεί, Πρόεδρε, είναι ότι το κοινοβούλιο αυτό κατανοητά είναι διχασμένο και ότι η επιρροή του Ισραήλ είναι τέτοια που θα προσπαθήσει να πνίξει κάθε σχετική συζήτηση. Είναι λοιπόν κρίσιμη σημασία στο Ισραήλ να λάβει επιβεβαίωση για την ύπαρξή του, για το μέλλον του, για τα σύνορά του. Αυτό είναι αυτονόητο και θα πρέπει να το επαναλαμβάνουμε. Αλλά είναι εξίσου αυτονόητο ότι και οι Παλαιστίνοι θα πρέπει να λάβουν μια διαβεβαίωση ότι έχουν και αυτοί μέλλον. Και αυτοί τους οποίους συνάντησα από το Χαμάς, από τη Χαμάς, μου φαίνεται ότι είναι πολύ αξιοσημείωτα άτομα με πολύ σαφή ιδέα για το τι θέλουν να πετύχουν πολιτικό πώς. Και τώρα ενώνονται με τη Φατάχ και θεωρώ ότι οι ελπίδες όλων μας που ενδιαφερόμαστε για το θέμα αυτό θα ενισχυθούν. Το Ισραήλ όμως θα πρέπει να πιεστεί τώρα για να καταλάβει ότι αυτά που λέει ο Ομπάμα θα πραγματοποιηθούν. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι τα σύνορά τους είναι ασφαλή, αλλά θα πρέπει να σταματήσουν οι επικισμοί, θα πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος η Γάζα, θα πρέπει να λάβει το καθεστώς που χρειάζεται και θα πρέπει να υπάρξει ελευθερία κίνησης για όλους τους Παλαιστινίους. Οι διπλωμάτες της Νοτιοαφρικής μου είπαν την τελευταία φορά που βρέθηκα εκεί, αν θεωρείτε ότι ο Απαρτχάιτ ήταν κακό στην Αφρική, ελάτε εδώ να δείτε με τα ίδια στα μάτια σας τι, σημαίνει, τι συμβαίνει. Αυτό είναι πραγματικά θλιβερό και θα πρέπει να το έχουμε υπόψη όταν κάνουμε τι συζητήσεις αυτέ. Και τέλο, Πρόεδρε, θα πρέπει να γίνει μια μεγάλη συζήτηση με θετικά αποτελέσματα, ειδικέ, συγκεκριμένε πολιτικέ που πρόκειται να προωθήσουμε. Είτε πρόκειται για το εμπόριο, την πολιτική, την οικονομία, θα πρέπει να είμαστε πλέον μεγάλοι παράγοντες και όχι απλά να πληρώνουμε. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη ευκαιρία την οποία δεν πρέπει να χάσουμε. Ευχαριστώ. ένα από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ. Ήμουν και εγώ στην αντιπροσωπεία. Είμαι και αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας μάλιστα. Της αντιπροσωπείας με την Παλαιστίνη. Συμφωνώ απόλυτα με όσα είπε ο πρόεδρος Ντερόσα. Η ΕΠΑ πίεζε το Συνφέιν να πάει στις διαπραγματεύσεις. Ε, τότε ήταν τρομοκράτες. Ήταν λίγο πιο προσεκτικές πάντων. Επειδή είπατε κάτι για τρομοκράτες κύριε Ντερόσα, ε, το σκέφτηκα. Το Συμβούλιο και η κυρία Άστον. Το ψήφισμα των είναι καλό, αλλά τι λέμε, όταν λέμε ότι όταν είναι κατάλληλο ο χρόνο, τι εννοούμε στο άρθρο 2. Αυτό που εμείς λέμε ή εσείς λέτε ειρηνευτική διαδικασία ουσιαστικά παρατείνει και διευκολύνει την κατοχή. Η κατοχή έχει συνεχιστεί, συνεχίζεται, συνεχίζεται και λαμβάνονται μονομερή μέτρα από το Ισραήλ οι επικισμοί είναι σίγουρα ένα μονομερές μέτρο. Το τείχος είναι μονομερές μέτρο. Η παρέτσα θέλετε για την για τη γάζ. Πάλι είναι μονομερές. Άρα, καλό θα ήταν να βλέπουμε να κάνουν και δύο πλευρές πράγματα. Πρέπει να έχουμε όμως το εξή. Τα δικαιώματα δεν είναι υποσυζήτηση. Δικαιώματα υπάρχουν. Είναι σαφή. Σύνορα και τα λοιπά βάσει του διεθνούς δικαίου. Πρέπει να σταματήσει η κατοχή και μετά να συζητήσουμε και να διαπραγματευτούμε τους πρόσφυγε τι θα κάνουμε, πώς θα τα κάνουμε κτλ. Δύο κυρίαρχα κράτη θα είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τελευταία παρατήρηση. Ο χρόνος εξαντλείται. Πραγματικά εξαντλείται. Και θα ήταν τραγική λύση του ενός κράτους. Έχω συναντηθεί με πολλούς Παλαιστινίους που πιστεύουν ότι μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Γιατί λένε ότι ίσως για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση ανταποκριθεί στις ε, υποχρεώσεις της και μιλήσει για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι σωστό αυτό, αλλά εγώ νομίζω ότι θα έχουμε δεκαετίες μίσους και βίας. Θα έχουμε πραγματικά πολλούς θανάτους αν χρειαστεί να παραιτηθούν από τη λύση των δύο κρατών. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει παραμικρή πρόοδος. Θα δεχθούμε αυτό που λέει ε, η Επιτροπή Θα πετάξουμε στα σκουπίδια το μόνο καλό που υπάρχει. Νομίζω ότι η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πληγεί πάρα πολύ σε ολόκληρη την περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή. Ehm. Ευχαριστώ για όνομα αντιπαθείς γιατί πρέπει να σας θυμίσω συνέχεια το χρόνο. Δυστυχώς, παρότι θέλουν πολλοί συνάδελφοι, πέντε τον αριθμό, να παρέμβουν και άλλοι πολλοί, αλλά τέλο πάντων πέντε έχω γραμμένους εγώ, θα απαντήσει σε σύντομα και ο κύριος Ντερόσα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σύντομα παρακαλώ λοιπόν όλοι, ο κύριος Μπρόκ. Πρόεδρε, κάποιε σύντομε παρατηρήσει. Να θέσω το αγαπημένο μου ερώτημα πότε θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο κουαρτέτο να αναλάβει σημαντικό ρόλο έναντι των ΙΠΑ ε, και να μην ε, υιοθετεί πάντα το ρόλο, το βοηθητικό. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό ερώτημα και σε ό,τι αφορά την επίλυση των ε, προβλημάτων στην περιοχή. Νομίζω ότι αν η Ευρώπη και οι ΗΠΑ αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην περιοχή αυτή θα υπάρξει η απαραίτητη ασφάλεια, η απαραίτητη εμπιστοσύνη στην διαδικασία αυτή. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει λοιπόν ε, να διευκρινίσουμε ότι αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες αποτελούν το πρόβλημα. Μπορούμε να ζητάμε για ποιους λόγους η Χαμάς ε, έχει διαμορφωθεί όπως έχει διαμορφωθεί στη Γάσα. Μπορεί να μπορούμε να διαφωνούμε για τους λόγους αυτούς, αλλά όσο υπάρχει ισχυρή δύναμη από πολυεθνικής πλευράς και αρνείται να αναγνωρίσει την ε, ύπαρξη του Ισραηλινού κράτους, έχουμε και από τις δύο πλευρές ένα πρόβλημα πέρα από την κριτική για την ε, πολιτική επικισμού του Ισραήλ, θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό, το οποίο ασφαλώς αποτελεί εξίσου σημαντικό πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε να υπάρξει μια διαδικασία η οποία θα απολαμβάνει την υποστήριξη και των δύο πλευρών. Αν θέλουμε να υπάρξει συμφωνία των δύο πλευρών, αν η διαδικασία αυτή δεν θέλουμε να καταδικαστεί. Και θα πρέπει θεωρώ στη συνέχεια, σε συνεργασία με τον Αραβικό Σύνδεσμο και με τα άλλα αραβικά κράτη, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Να δούμε πού μπορούν να συνεχιστούν οι δημοκρατικές ε, εξελίξεις. Αλλά αυτό θα έχει συνέπειες και σε ό,τι αφορά το Ισραήλ. Ε, συνέπειες που δεν μπορούμε να ξέρουμε ούτε εμείς ούτε το Ισραήλ και γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί αυτό το ζήτημα. Θεωρώ ότι η επίλυση του Μεσανατολικού είναι κάτι που αποτελεί επιτακτική ανάγκη αν θέλουμε ειρήνη στο σύνολο της ε, περιοχής αυτής. Ευχαριστώ. Κολέγα Κιλ Νίλσεν, παρόλα. Κιλ Νίλσεν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε μου δίνετε το λόγο. Πράγματι μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι είναι εξαιρετική η του κυρίου Ντερόσα. Πρέπει να γίνει συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Το βλέπουμε αυτό. Απαιτεί το όλο θέμα μία μακρά συζήτηση, άρα συμφωνώ με την πρόταση αυτή. Θα ήθελα να επανέλθω σε κάποιε από τι παρατηρήσει που έγιναν. Πρώτα απ' όλα, λέει ο κύριο Μπροκ, πρέπει να ρυθμίσουμε το θέμα για την ε, περιοχή. Όχι κύριε Μπροκ, είναι σημαντικό για όλους, για τις δικές μας πόλεις, για την ε, σταθερότητα, ε, την ηρεμία και στις δικές μας τις πόλεις και στις δικές μας χώρες. Να επανέλθω σε μια φράση που ακούστηκε πριν, ότι ε, κινδυνεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση να χάσει την αξιοπιστία της. Λυπούμε, αλλά φοβάμαι ότι ήδη συμβαίνει αυτό. Αν δει κανείς ότι η κοινωνία των πολιτών ε, παίρνει ε, την κατάσταση στα χέρια της, γιατί εμείς δεν κάνουμε τη δουλειά μας. Όταν βλέπουμε αυτή την εκστρατεία μποϊκοτάζ των επενδύσεων ε, για τον αποκλεισμό προϊόντων από τις απικίες, κάτι που βλέπουμε σε πολλές χώρες, επειδή δεν μπορεί η Γαλλία να ε, εξασφαλίσει τη σωστή ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, στο πλαίσιο με το Ισραήλ. Δεν γίνεται σεβαστό το διεθνές δίκαιο, η σύμβαση της ε, Γενέβης. Λοιπόν, εδώ έχουμε απογοήτευση και αποστασιοποίηση από τους πολίτες. Ε, το βλέπουμε και με τη Γάζα. Ο αποκλεισμό της Γάζας είναι απαράδεκτο. Όπως και άλλοι συνάδελφοι, και εγώ έχω μεταβεί στη Γάζα Πλιστάκη. Ο αποκλεισμό τη Γάζας από ανθρωπιστική πλευρά είναι απαράδεκτος. Πάνω από το 60% του πληθυσμού είναι ανήλικοι, είναι παιδιά, τα οποία πληρώνουν το τίμημα κάποιων που το 2006 ε, έκαναν ε, στις εκλογές κάτι που δεν μας άρεσε, ψήφισαν προς τη λάθος κατεύθυνση. Λοιπόν, ε, είναι απαράδεκτο για την νεολαία αυτό και πάρα πολύ επικίνδυνο. Και θέλω να πω κάτι απλό. Ο Στολίσκος, για τον οποίο έγινε λόγο πέρυσι. Ίσως έκανε το Ισραήλ να αντιδράσει για κάποιο χρόνο, γιατί κάπως ελάφρυναν τον αποκλεισμό, αλλά καθόλου δεν είναι αυτό ικανοποιητικό, είναι θα έλεγα μία αυταπάτη. 15 πλοία αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται ε, να καταπλέψουν προς τη Γάζα. Προέρχονται από πολλές χώρες της Ευρώπης. Στη Γαλλία το πλοίο για την Ειρήνη, το πλοίο για τη Γάζα ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή έχει μια εξαιρετική στήριξη από το λαό της χώρας μας. Ε, δημοσιογράφοι, όχι μόνο πολιτικοί και άλλοι εκτός του πολιτικού κόσμου, στηρίζουν αυτό το στόλο για τη Γάζα και πραγματικά ελπίζω κυρία Άστον και η υπηρεσία της να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο σε επαφές με τις Ισραηλινές αρχές για να μην έχουμε όπως την προηγούμενη χρονιά αυτή την επίθεση των ε, φιλιρινικών διαδηλωτών που κατευθύνονται προς τη Γάζη για να καταγγείλουν τον αποκλεισμό και να μην έχουμε αιματοχυσία. Ευχαριστώ. Κυρία Γκόμες, να σας πω ότι πρέπει να περιοριστείτε σε ένα λεπτό, ένα μισή λεπτό, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ιδάλλως άλλωστε θα έχουμε χρόνο για τους υπόλοιπους συναδέλφους. Ναι, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να υποστηρίξω την ιδέα αυτή της ε, διοργάνωσης μιας συζήτησης με τη συμμετοχή της κυρίας Άστον. Προκειμένου να τοποθετηθεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεωρώ ότι είναι πραγματικά κρίσιμη η χρονική συγκυρία. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αυτό το αδιέξοδο. Η Αραβική Άνοιξη έχει αλλάξει την κατάσταση για το Ισραήλ. Το, θέμα δεν είναι το Ισραήλ τώρα, αλλά θα είναι στο μέλλον αν δεν συμβεί τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν οπωσδήποτε θα πρέπει να τοποθετηθεί, να τοποθετηθεί το Κοινοβούλιο, να απαιτήσει από το Συμβούλιο να ηγηθεί. Το θέμα δεν είναι να είμαστε ίσοι με τη ΣΥΠΑ, όχι. Το θέμα είναι να κάνουμε ό,τι κάναν όταν ενέκριναν την ε, δήλωση της Νίκαιας. Και θέλουμε να το κάνουμε αυτό και το θέμα αυτό αφορά την ασφάλειά μας, όπως και το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Thank you. Noiser, ε, ε, please. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ήμουν και εγώ, συμμετείχα και εγώ στην αποστολή αυτή θα μπορούσα πολλές λεπτομέρειες να σας παρουσιάσω που καταστούν σαφές ότι η εκδίωξη έχει γίνει ακόμα πιο βίαιη, που καταστούν σαφές ότι η ανθρωπιστική κατάσταση έχει επιδεινωθεί περαιτέρω. Νομίζω ότι η ανεξάρτητη έκθεση του ΟΗΕ αποτελεί σαφές τεκμήριο όλων αυτών και πιστεύω ότι σήμερα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει δεν έχω όρεξη να κάθομαι πάντα ως βουλευτής και να σκεφτόμαι κατά πόσο θα πρέπει να αναλάβει δράση το Συμβούλιο. Όχι, θα πρέπει να παίξουμε το ρόλο μας και θα πρέπει να τοποθετηθούμε με σαφήνεια και μάλιστα εγκαίρως ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Σεπτέμβριο θα υπάρξει, θα ληφθεί η απόφαση για τον ΟΗΕ και θα πρέπει να έχει λάβει μέχρι τότε θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αλλιώς θα χάσουμε κάθε ευκαιρία αξιοπιστίας έναντι του αραβικού κόσμου όταν ε, διεξάγεται μια τέτοια διαδικασία και εμείς δεν τοποθετούμαστε με σαφήνεια. Ευχαριστώ. Τελευταίος ο μελητής. Ευχαριστώ. Επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, θα ήθελα να ζητήσω, να θέσω μία ερώτηση η εκπρόσωπο τη Υπηρεσία Εξωτερικής Δράση, της κυρία Άστον ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή οι ευρωπαϊκοί φορολογούμενοι πληρώνουν 500 εκατομμύρια το χρόνο ως βοήθεια για τους Παλαιστινίους. Ερωτώ, το κράτος του Ισραήλ έχει πληρώσει αποζημίωση για όσες ε, ζημίες έχει προκαλέσει το κράτος του Ισραήλ και έχει ζητήσει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση από το κράτος του Ισραήλ να, να πληρώσει αποζημίωση για τις παραβιάσεις διεθνούς δικαίου που έχει διαπράξει. Για παράδειγμα, την παράνομη επίθεση στη Γάζα. Ή μήπως υπάρχει κάποιος κανόνας ότι οι Ευρωπαίοι δάσκαλοι και οι προσβέστε πρέπει να πληρώνουν για να ξαναφτιάχνονται τα κτίρια που έχουν καταστρέψει οι Ισραηλοί. Λοιπόν, πολύ σύντομα τα συμπεράσματα, δύο λεπτά. Άντε, δυόμιση λεπτά. Στον κύριο Ντερόσα και στην κυρία Σμιτ. Η κυρία Σμιτ πρώτα και μετά ο κύριος Ντερόσα. Πολύ σύντομα γιατί πρέπει να κλείσει η σημερινή συνάντηση. Α, είμαι πάρα πολύ σύντομη για την ερώτηση του κυρίου Μπροκ για το πότε θα αναλάβουμε τον ηγετικό μας ρόλο. Το κουαρτέτο περιλαμβάνει τέσσερα μέλη, την ΣΥΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ρωσία και τον ΟΗΕ. Αυτό έχει να κάνει και με το που συναντιέται το κουαρτέτο, για το ποιο δηλαδή έχει την ηγετική θέση. Η δάλος είναι σαφής οι σχέσεις και οι αναλογίες και αυτό ήταν σαφές ήδη από το 2002. Το θέμα είναι θέμα εφαρμογής και νομίζω ότι εμείς έχουμε το βασικό ρόλο. Θα πρέπει να βρεθεί λύση και θεωρούμε θεωρώ ότι θα πρέπει να, υπάρχουν, να υπάρχει συμμετοχή και των δύο μερών. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με μονομερή βήματα. Θα πρέπει επίσης να πω ότι το Ισραήλ επί μεγάλο χρονικό διάστημα να μην ξεχνάμε και τις διαδικασίες και τις επιθέσεις στη Γάζα. Αυτό ίσως είναι κάτι που το τίνουμε να το ξεχνάμε. Yeah, uh, συμπέρασμα λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ για να αποφύγουμε μακροσκελή σχόλια σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις της Ισραηλινές. Χορηγήθηκαν αποζημιώσεις στον ΟΗΕ για υποδομές που καταστρέφηκαν στην Γάζα. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αποζημιωθεί, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί τις ε, υποδομές αυτές στους Παλαιστινίους. Οι Παλαιστίνοι λοιπόν θα έπρεπε να ζητήσουν ενδεχομένω αποζημίωση για τα συστήματα αυτά. Για το θέμα της Χαμάς, να απαντήσω. Η Χαμάς, όπως όλες οι οργανώσεις που προκύπτουν από αγώνες απελευθέρωσης, περιλαμβάνει πολιτικούς, τρομοκράτες, άτομα που κινούνται μεταξύ των δύο αυτών στρατοπέδων αποτελεί ένα κίνημα το οποίο εξελίσσεται. Το γεγονός ότι α, σύναψαν αυτή τη συμφωνία η ειρηνευτική διαδικασία αποτελεί τεκμήριο του γεγονότος αυτού. Δεν λέμε ότι απαραίτητα θα πρέπει να υπάρξει συμβιβασμό, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση για να αναπτυχθεί η γλώσσα που είναι απαραίτητη προκειμένου να λάβει τις διαβεβαιώσεις που χρειάζεται το Ισραήλ. Ιδάλλως, δεν είμαστε σοβαροί. Αν δεν δεσμευτούμε, δεν επιδεικνύουμε σοβαρότητα. Και αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να το έχουμε υπόψη. Επίσης να πω ότι ε, υποστηρίζω απόλυτα την δήλωση του α, Συμβουλίου για τον Σαλής, ο οποίος θα πρέπει να απελευθερωθεί. Αλλά θα ήθελα το Συμβούλιο να πει μια φορά ότι τα 600 παιδιά της Παλαιστίνης που κρατούνται σε φυλακές και αυτά θα πρέπει επιτέλους να απελευθερωθούν. Θα πρέπει να είναι ε, ισόρροπη η προσέγγιση που θα ακολουθήσουμε. Καταλαβαίνω ότι ο Σαλής θα πρέπει να επιστρέψει στην οικογένειά του, αλλά οι ανθρωπιστικές ανησυχίες θα πρέπει να αφορούν όλες τις πλευρές. Και περνάμε και μιλάμε για παιδιά τα οποία θα πρέπει να περάσουν από δικείο και αυτά θα πρέπει να απελευθερωθούν. Ωραία, σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας, για την παρουσία σας. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9.